Καλημέρα σα. Αρχίζουμε σήμερα με ψηφοφορία την έκθεση συναδέλφου Κουρία Αναγνώριση και Προώθηση Διασυνοριακών Εθελοντικών Δραστηριοτήτων στην Ένωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ντόρις. Να ευχαριστήσω την γραμματεία, τον κύριο Φοντανίλη. Επίσης, να τονίσω και την αρμονική συνεργασία με τους κεώδεις εισηγητές. Ήταν πραγματικά δουλειά ομάδας, όπως ο εθελοντισμός διδάσκει. Ευχαριστώ. Περνούμε λοιπόν αμέσως στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Πιστεύω. Εντάξει, πάμε. Η τροπολογία παριθμών 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 10. 11. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 είπε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 είπε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 είπε, Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την 39. Πέρας. 11-12 απορρίπτεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. 12 ναι, εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 46 έχει αποσυρθεί. Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα μάλλον. 47 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχής ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 15-8 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Αρχίζει η ψηφοφορία για την 69. 1214 απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος. Αρχίζει ψηφοφορία. Τελειώνει αμέσω. 11-14 απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 79 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 78 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 80 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχή ψηφοφορία. Τελειώνει αμέσω. Απορρίπτεται 10-16. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ ορίστε 88 έκανα λάθος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 14-13 εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Αυτό τώρα τι είναι. Υπέρ είσαι. Μάρκο, είσαι κατά του συμβιβασμού. Δεν ψηφίζεις. Α, in favor, ωραία. Ε, γιατί τρόμαξα. Συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει προφορία για τη συμβαστική 5. Πέρας. 18-9 εγκρίνεται. 104. Ψήφι υπέρ. Κατά Υπέρ είστε, εντάξει, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική 2 εισηγητής υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 9 προς 13 και 5 εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά ξανά 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα που πάμε Στη 14, είπε κατα Κατά. Εποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχής προφορία. Τελειώνει. Απορρίπτεται 11-16. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές ξανά. Την 20 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Α, ισοψηφία απορρίπτεται. Τι να κάνουμε έτσι έχει η ζωή. 21 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 είπε. κατα Κατά αποχές έλεγχος. Αρχής Περάσα. 15-13 εγκρίνεται. 23 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, έχω να σας κάνω την εξής πρόταση. Έχει παντού θετικό πρόσημο και για τον εισηγητή για όλες τις τροπολογίες της ε, απασχόλησης.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 Αρχίζω τραγουδάω, λέει η 17 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι, όχι, ανέκδοτο ήταν. Πλάκα έκανα, ναι. Λοιπόν, 16 <laughs> υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 26 υπέρ με 2 αποχές και 0 ψήφους κατά. Ήταν πρωινή γυμναστική αυτή, εντάξει. Μερικοί όμω δεν είχαν γυμναστική και πρέπει να μυρίζουν τα νύχια μου για να καταλάβω τι θέλετε. Λοιπόν, τελειώνει εδώ η πληροφορία. Ελπίζω να παραμείνουν μερικοί και να μην εξαφανιστούν τρέχοντας. Η κυρία Παλιαδέλη. Κυρία Παλιαδέλη. Κυρία Παλιαδέλη, πού πάτε. Ε, προσβλέπαμε στην ε, παρουσία σας. It was, I was joking. So, we, Λοιπόν, ακρόαση έχουμε τώρα. για το μελλοντικό πρόγραμμα πολιτισμού, ε, μέσων ε, ενημέρωσης και του κλάδου της δημιουργικής οικονομικού κλάδου της δημιουργίας. Λοιπόν, αν θέλετε να βγείτε, ε, αποχωρήστε ησύχως τουλάχιστον και να μην κάνετε φασαρία και ενοχλείτε τη συνεδρίαση. Στο καλό, γεια σας. Χαίρομαι που έχουμε φέρει εδώ εμπειρογνώμονες. Έχουμε τον κύριο Βαλέριο Καρούσο, διευθυντή του ΣΥΝΟΕΡΟΠΑ, εδώ μπροστά κάθεται. Καλωσορίζουμε τον κύριο Όλαφ Τσίμερμαν, Διευθυντή ε, του Γερμανικού ε, Πολιτιστικού Συμβουλίου. Έχουμε τον καθηγητή Ντάβιτ Χεσμοντάλκ, που είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου ε, Επιστημών Επικοινωνίας και καθηγητής Μίδια και Μουσικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο του Λίτς και τον κύριο Ράντου Μιχαλιάνου, ο οποίος είναι σκηνοθέτης επίτιμος πρόεδρος ε, της Επιτροπής για το βραβείο Λουξ φέτος. Πού είναι? Α, θα είναι καθοδόν. Äh, λοιπόν, να σας πω πώς θα το οργανώσουμε. Θα... Κάθε πυρογνώμο 10 λεπτά και μετά οι συνάδελφοι. Και μετά θα έχουμε πάλι την ευκαιρία 5-10 λεπτά να ακούσουμε απαντήσεις των ειδικών μας και βεβαίω θα δώσω λόγο και στην Προεδρία του Συμβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουν σχόλια. Ο κύριος Χανσίστιαν Κρίστενσεν εκπροσωπεί το Συμβούλιο και τη Δανική Προεδρία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Διευθυντής για τον Πολιτισμό και τα Μίδια, ο κύριος Βλαντιμίρ Σούχα. θα πρέπει να συζητήσουμε το νέο πρόγραμμα, ε, ενδεχομένω να το τροποποιήσουμε και κάποια στιγμή να το εγκρίνουμε κιόλα. Έχει άλλο όνομα από ό,τι στο παρελθόν. Έχει να κάνει με τον πολιτισμό και το ε, οικονομικό κλάδο της δημιουργίας. Βέβαια το σημαντικό πρόγραμμα Media που ήταν τόσο σημαντικό για μας δεν εξαφανίζεται, παραμένει, έχει αλλάξει ο τίτλος. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Προβλήματα έχουμε σίγουρα με το θέμα, τον όρο στα αγγλικά Creative Industries. Γνωρίζετε όλοι πόσο μικρός είναι ο προπολογισμό και γι' αυτό μας απασχολεί ακριβώς πώς μπορούμε να επηρεάσουμε κάπως αυτό το κλάδο της ε, δημιουργίας και που είναι ε, οι ε, πολιτιστικές πρωτοβουλίες περιφερειακής ε, διάστασης που παίζουν πολύ μεγάλη πολύ μεγάλο ρόλο συγγνώμη, στη ζωή μας. Γίνονται συζητήσεις πολλές σε πολλά κράτη-μέλη, πολλές είναι οι αγωνίες και οι φόβοι και η σημερινή ακρόαση θα μας δείξει λίγο ποιο είναι τώρα το στάδιο της κατάστασης, ποια είναι τα θέματα που διαπραγματεύεται, ποιε είναι οι αγωνίε και οι φόβοι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούν αυτά να διασκεδαστούν. Και χτες ακούσαμε για άλλο πρόγραμμα ότι ήθελαν να μας καθησυχάσουν. Και είπα, δεν θέλω να με καθησυχάσετε. Θέλω από την αρχή να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για να μην χρειάζεται να ανησυχήσω και να με καθησυχάσετε. Γι' αυτό ελπίζω σήμερα ορισμένε αγωνίες να τις καταρρύψουμε και να τις ξεπεράσουμε και να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα. Και τελικά να έχουμε το πρόγραμμα που χρειαζόμαστε και που επιθυμούμε όλοι. Γιατί έχουμε καλή εμπειρία με το πρόγραμμα. Nicht überlagert wird και ελπίζω να μην ε, το υπερφορτώσουν και να μην ε, επισκιαστεί από τα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί τα συμφέροντα του πολιτισμού δεν είναι πάντα οικονομικά, αλλά έχουν και άλλο χαρακτήρα. Λοιπόν, να σταματήσω εγώ εδώ την εισαγωγή μου και να δώσω το λόγο στον πρώτο εμπειρογνώμονα και χαίρομαι που ο κύριος Καρούσο θα πάρει το λόγο για 5-10 λεπτά ή 15 λεπτά αν θέλει. Είναι ο επικεφαλής ε, του ΣΥΝ Ρόπα που μας βοηθάει πάρα πολύ ε, και στο βραβείο Λουξ και τους 27 νέους που καλούμε στη Βενετία για τις μέρες της Βενετίας ε, με αφορμή το βραβείο Λουξ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ κυρία Πακ, ευχαριστώ και την Επιτροπή Πολιτισμού που με κάλεσε. μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι. Πριν ξεκινήσω να πω ότι πρόκειται για μια ε, μεγάλη ευθύνη να παρουσιάζει κανείς ε, τις προοπτικές του Μέντια και του Μέντια Μούντους. Εγώ διαβουλεύθηκα με πολλές ε, οργανώσεις, χωρίς να είμαι εκπρόσωπός τους, θα κοιτάξω να σας δώσω μία περίληψη των πιο ενδιαφερουσών προτάσεων που προέκυψαν από την συνεργασία μου με αυτές τις οργανώσεις. Τώρα πριν να ξεκινήσω να σας αναφέρω εδώ μερικά στοιχεία τα οποία ανατρέπουν εντελώς την κατανάλωση και διανομή των έργων στο μέλλον. Πέρα ε, το 2013 θα έχουμε 3,4 δις καταναλωτών στο ίντερνετ ε, καταναλωτές επίσης ε, κινητών ψηφιακών ταμπλετών, ε, iPhone, iPad κλπ. Τρία δισεκατομμύρια τέτοια μηχανάκια που έχουν πολιθεί ανά τον κόσμο. Και αυτή η υποδομή χρησιμοποιείται και για την προβολή τένιων Δηλαδή, ο όρος smart θα αποτελέσει επίκεντρο της ζωής μας, είτε smartphone, είτε smart οτιδήποτε συνδέεται στο ίντερνετ. Και η φυσική βάση θα εξαφανιστεί στο μέλλον. Θα υπάρχει ένας, θα, θα υπάρχει ένας χώρος όπου θα αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία έξω από το υπολογιστή στο σπίτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ένα φιλμ στο smartphone, μπορούμε και μετά να το περάσουμε στο iPad και μετά στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το ίντερνετ. Πρόκειται για το σχέδιο κοσμέρια, δηλαδή το οπτικακουστικό προϊόν διαχωρίζεται σε πολλές θεματικές. Μπορούμε να έχουμε μια ταινία μεγάλου μήκους 80 λεπτών που να γίνεται ε, ε μίνι σειρά των 10 λεπτών στο τηλέφωνο και ε, να, είναι, και να σπάζει σε άλλα κομμάτια για το iPad. Εδώ βλέπετε ποιες είναι οι προσφορές video on demand και συνδρομητές στο video on demand ε, τα τελευταία χρόνια και ποιες είναι οι προπτικές για το 2016. Το 2011 τα DVD και τα Blu-ray ε, που λιόντουσαν στο ίντερνετ, σήμερα όμως αυτό θα αλλάξει. θα έχουμε τρία δις πωλήσει online έναντι των δύο δις ε, ε, υλικών πωλήσεων. Σε 10 χρόνια έχουμε μία σημαντική αύξηση των πωλήσεων online. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Καταρχήν κατακαιρματισμός της ακροματικότητας. Όποιος ε, μιλάει για πέρασμα της ακροματικότητας ε, προς το ίντερνετ σημαίνει μείωση ακρωματικότητας της τηλεόρασης, αυτό σημαίνει μείωση των διαφημιστικών εσόδων και μείωση των παραγωγών, των τηλεοπτικών παραγωγών. Ήδη η παραγωγή DVD και Blu-ray είχε μειώσει τα έσοδα των ε, παραγωγών και είναι ανησυχητικό αυτό το, ε, αυτό, αυτό, αυτό το στοιχείο. Στις Ηνωμένε Πολιτείες οφείλεται αυτό στην δυνατότητα συνδρομής σε βίντεο on demand στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δηλαδή, ε, μέσα από μία καταποκοπή συνδρομή ε, κάθε μήνα, μπορεί κανείς να βλέπει ένα συγκεκριμένο οπτικακουστικό ε, πρόγραμμα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, ε, το 94, το, ένα μεγάλο ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά καλύπτεται από αυτού του είδους την συνδρομή. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, το να δει κανείς μια ταινία στοιχίζει 51 cent με SVOD. Ενώ αν αγοράσει το DVD στοιχίζει 4,72 δολάρια. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τους νέους ε, γίγαντες της ε, διανομής που είναι η Apple, η Netflix, η Google Play και η Amazon που θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Τώρα για να μπούμε πραγματικά στο ψητό, δηλαδή το πρόγραμμα Μέντια, είναι φανερό ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έλαβαν υπόψη τους όλες αυτές τις αλλαγές με τους νέους λειτουργούς που μπαίνουν στην αγορά και είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς και τους διανομείς στην Ευρώπη να δούνε πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτόν τον νέο τρόπο ε, θέασης ε, του οπτικακουστικού μέσου. Τώρα έχουμε ένα νέο λάμπελ, μια ποιότητα ένα σήμα ποιότητας ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες με σαφείς ε, κατευθυντήριες γραμμές με ένα αποτελεσματικό ε, σύστημα ε, ε, πληρωμής. Το σύστημα των media δημιούργησε ένα στενό δεσμό με τους λειτουργούς του οπτικακουστικού. Ας δώσουμε λοιπόν μια καλή εικόνα της Ευρώπης προς τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεδομένων των αλλαγών που θα υπάρξουν στην αγορά των οπτικακουστικών, δεν θα πρέπει να υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού στο πρόγραμμα Μέντια διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδεύσει όλες αυτές τις αλλαγές. Πιστεύω, όπως και πολλές άλλες οργανώσεις στην Ευρώπη, ότι μέσα στο πακέτο της Creative Europe να υπάρχει μία σαφής, ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ των μίδια και του πολιτισμού και του προγράμματος αυτού καθεαυτού το πρόγραμμα Media πρέπει να είναι διαπιστώσιμο. Τώρα για τα Media Desk και τα γραφεία πληροφόρησης για τον πολιτισμό θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ καλή ιδέα για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ένα κόστος, αλλά αναρωτιέμαι ε, αν η εμπειρία αυτών των δύο δικτύων τελικά χαθεί. Εμείς επίσης βλέπουμε πολύ θετικά αυτά τα πολυετή συμβόλαια που θα ευνοήσουν και τους δικιούχους αλλά και τον οργανισμό που διαχειρίζεται τα συμβόλαια. Πρέπει να μπούμε σε μια προοπτική συνέχεια με αυτά τα οποία έχουμε κάνει με τα προηγούμενα προγράμματα και να υποστηρίξουμε τους ίδιους τομείς που υποστηρίζαμε και στο παρελθόν. Με ένα νέο ε, κεφάλαιο τα ε, media Τώρα για τους τομείς ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιήσει ο επαγγελματίας την άφηξη των νέων τεχνολογιών, να ορίσουμε το νομικό πλαίσιο που θα αλλάξει σε αυτήν τη νέα ψηφιακή εποχή και για την βοήθεια προς τους παραγωγούς, δηλαδή το κεφάλαιο που αφορά δηλαδή ε, την ανάπτυξη αλλά και τις ε, τηλεοπτικές μεταδόσεις. Αν δούμε το, ε, ε τις τελευταίες δημο... Τους τελευταίους ε, διαγωνισμούς ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σκαντανέβασμα και ως προς τις χώρες ε, αλλά και ως προς τους δικιούχους. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, να υποστηρίζουμε και τον τομέα των εφουσών κινηματογράφου που είναι σημαντικός για την θέαση των κινηματογραφικών ταινιών. Εάν δούμε τα στοιχεία του Europa Cinema, ε, εάν ε, βλέπουμε ότι έξι στις 10 προβολές ε, είναι ευρωπαϊκές και άμα βγάλουμε τον ε, Χάρι Πότερ ο οποίος είναι μεν βρετανικός αλλά με αμερικανικά λεφτά ε, το 35% είναι ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να ε, χρηματοδοτήσουμε πολλές ε, πλατφόρμες video on demand όταν ε, το μέγεθος της αγοράς δεν μας επιτρέπει να τις υποστηρίξουμε όλες. Μήπως θα έπρεπε να εργαστούμε για τη δημιουργία μίας ή δύο πλατφορμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπλέκοντας και τις τηλεοράσεις. Ξέρουμε ότι ε, οι τηλεοράσεις έχουν ενεπτυγμένο ε, δίκτυο ε, video on demand ή catch-up TV και μπορούν να το αναλάβουν. Τώρα ε, μπορούμε να είδαμε για το Teramento Plus ε, ότι όταν υπάρχει βούληση, πολιτική βούληση μπορούμε να βάλουμε μαζί τις τηλεοράσεις. Έχουμε έξι τηλεοράσεις ε, ε, οι οποίες ε, συνέπραξαν ε, πρόκειται για τέσσερα ευρωπαϊκά κανάλια και δύο μεσογειακά από την Αλγερία και το Μαρόκο και προσφέρουν βίντεο on demand σε αγγλικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα αραβικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε επίσης ε, και το θέμα ε, των εθουσών είπαμε κινηματογράφου. Πρέπει να συνεχίσουμε να να προωθούμε τις ε, ταινίε με τη δημιουργία πολύγλωσσων καναλιών. Αξίζει τον κόπο εκ μέρους ε, της Κομισιόν να καταβληθεί μία προσπάθεια για έναν καλύτερο ορισμό του δημοσιονομικού μέσου. Όταν εμείς ε, μιλάμε για το Ταμείο Εγγύσεων που είναι εξαιρετική πρωτοβουλία, θα έπρεπε να ψάξουμε να, να, δημιουργήσουμε περισσότερους ε, ε, χρήστες. Εμείς τώρα έχουμε τους ιστορικούς ε, χρήστες, θα έπρεπε να βρούμε και άλλους. Για το Media Mundus. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε το Media Mundus στο πρόγραμμα media, δηλαδή οι μη Ευρωπαίοι επαγγελματίε να μπορούν και αυτοί να έχουν πρόσβαση στα μέσα που προτείνει το media. Και για να τελειώνω, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε, όπως πάρα πολλές φορές το είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ε, μελλοντική, τη media literacy για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, μας δώσατε πολλές ιδέες, μερικές από αυτές ήταν και δικές μας ήδη. Η κυρία Κώστα που είναι η συγγήτρια θα τα καταγράψει όλα αυτά και τις ιδέες σας επίσης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Όλαφ Τσίμερμαν, Διευθυντή του Γερμανικού Πολιτιστικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν μας καλέσατε. Το Γερμανικό Πολιτιστικό Συμβούλιο είναι η οργάνωση που ε, συνενώνει 235 φορείς. Ε, είναι κάτι που αφορά όλους τους τομείς της τέχνης, μουσική, ε, φιλο λογία, οικαστικές τέχνες ε, και πολλά μέσα και ε, video games και παιχνίδια στους υπολογιστές. Είναι πολύ σημαντικό ότι πούμε στη Γερμανία την κοινωνία των πολιτών αλλά και τις δύο πλευρές αν θέλετε και τους καλλιτέχνες με τους συλλόγου και τις ενός τους αλλά και ε, τη βιομηχανία της δημιουργίας είναι και αυτή μέλη του, του Γερμανικού Πολιτιστικού Συμβουλίου όταν μιλούμε για την οργανωμένη κοινωνία πολιτών και τη συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών, καλύπτουμε ευρύ φάσμα συμφερόντων. Επιτρέψτε μου σήμερα να προσπαθήσω να αναφερθώ στα προγράμματα και της Δημιουργικής Ευρώπης από τη σκοπιά του πολιτισμού. Άκουσα ε, ότι οι συνάδελφοι είναι κυρίως από τα μίντια Και ε, εγώ θα προσπαθήσω περισσότερο από τον πολιτισμό για να ε, μην ε, υπάρξουν παρεξηγήσεις από την αρχή, για να μην έρχονται αντιμέτωπα αυτά τα δύο στοιχεία, πρέπει να σας πω ότι στη βιομηχανία της δημιουργίας πέρασα το μεγαλύτερο διάστημα του εργασιακού μου βίου. Δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. αν κοιτάξουμε αυτά τα προγράμματα θεωρούμε ότι είναι μονόπλευρα και γέρνει προς την πλευρά της βιομηχανίας της δημιουργίας. Το ξέρω ότι έχει σημασία, μας τα είπε ο κύριος Καρόζο θαυμάσια και δεν μπορώ παρά να το υποστηρίξω. Παρ' όλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι ένα πρόγραμμα που προωθεί και ενισχύει τον πολιτισμό δεν θα πρέπει να γίνει ε, ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του κλάδου, δηλαδή του οικονομικού της δημιουργίας. Μπορούμε να έχουμε προγράμματα διαρθρωτικά ή ειδικά οικονομικά που να στραφούν προς τα εκεί και όχι το πολιτιστικό πρόγραμμα. Στο σχέδιο προγράμματος που έχουμε θεωρούμε ότι η ίδια η αξία του πολιτισμού λαμβάνεται πολύ λίγο υπόψη. Δηλαδή η συνάντηση των πολιτισμών, πολιτιστική, η διαπολιτιστική πτυχή δεν έχει καλυφθεί επαρκώς και όλος ιδιαίτερος το όλο θέμα της εκπαίδευσης της πολιτιστικής δεν λαμβάνεται υπόψη όπως θα έπρεπε σήμερα να γίνεται. Η ιδέα είναι μια σύνδεση του προγράμματος για το πολιτισμό και του προγράμματος για τα μίντια. Το είπε και ο προλαλής σας. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα πολιτισμού και το πρόγραμμα μίντια είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι και τα δύο επιτυχημένα προγράμματα μέχρι σήμερα, τα οποία μπορεί κανείς έτσι να τα συνεχίσει αφού έχουν πετύχει. Τα πολιτιστικά προγράμματα στις διάφορες ε, τέχνες ε, έχουν ε, επιτύχει και έχουν προβληθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα πολιτιστικά προγράμματα ακριβώς ποντάρουν στην κινητικότητα των καλλιτεχνών, το να συναντώνται μεταξύ τους οι καλλιτέχνες πέρα από τα σύνορα, να διαδίδονται τα έργα τέχνης. Αυτό είναι και ο πυρήνας άλλωστε του προγράμματος για τον πολιτισμό. Και απευθύνονται σε ένα ευρύτατο κοινό. Αυτό το θεωρούμε πολύ θετικό. Και αυτό το κοινό, η ομάδα στόχος όπως ονομάζεται, ε, ε, δέχεται συμβουλές από διάφορα σημεία επαφής ε, στις διάφορες χώρες μέλη. Το να συνενωθούν τώρα τα δύο προγράμματα δεν το θεωρούμε πλέον έκτημα και δεν βλέπουμε ποιο είναι το καλό, για ποιο λόγο και ποια είναι η συνέργεια αν συνενωθούν αυτά τα δύο προγράμματα, αν συγχωνευτεί ο πολιτισμός με τα μέσα επικοινωνίας. Ίσως το μόνο πλεονέκτημα που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ότι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες καθοδήγησης και ε, για να περάσει μια γραμμή ε, πολιτιστική και πολιτική στα προγράμματα. Θα έρθω στη συνέχεια. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο, το ανέφερε και ο προλαλής σας, ήταν μεγάλη σπαζοκεφαλιά για μας που ασχοληθήκαμε με αυτό, διότι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ τον τρόπο λειτουργίας. Στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί. Περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα πρόγραμμα πιστώσεων, είναι ένα πρόγραμμα εγγύσεων, είναι ένα πρόγραμμα ενισχύσεων. Τι είναι. Δεν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να το απορρίψουμε ε, καταρχήν. Αλλά αν ενδιαφέρονται οι βουλευτές τουλάχιστον να προσπαθήσουμε εμείς να ελέγξουμε στις διάφορους τομείς της τέχνης πώς το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι επιπτώσεις θα είχε. Γιατί υπάρχει χρόνος, αν θέλετε να γίνει αυτός ο έλεγχος. Ακόμα και τώρα για μας ιδιαίτερο ρόλο παίζει η ενίσχυση των δικτύων. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, η ανάπτυξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στον πολιτισμό στην Ευρώπη. Και βέβαια το σχέδιο του προγράμματος αναφέρεται σε αυτό και θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχει η δυνατότητα της δικτύωσης και της χρηματοδότησης των δικτύων των πολιτών. Αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να γίνει περισσότερη αναφορά σε αυτό, έτσι ώστε οι διάφορες κοινωνίες των πολιτών στον πληθυντικό στην Ευρώπη που στα πολιτιστικά απέχουν μεταξύ τους πάρα πολύ και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να έρθουν πιο κοντά. Αυτοί λοιπόν χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα δίκτυο, μια υποδομή αξιόπιστη και φερέγγια. Και αυτό θα γίνει μόνο ε, στο διηνεκές και θα εξασφαλιστεί μόνο με θεσμική ενίσχυση και προώθηση. Και σας παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Προηγουμένως σας είπα ότι... να το πω αλλιώς. Έχω ένα αίτημα πιο ουσιαστικό και μπορεί να σας εκπλήξει που θα το ζητήσω εγώ ως Γερμανός. Κοιτάζοντας την εξέλιξη του προγράμματος και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα λέει το Συμβούλιο μας, πιστεύω ότι αυτή η κριτική μεταξύ άλλων προκύπτει και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι εμείς την αφήνουμε να κάνει, ό,τι εμείς της επιτρέπουμε να κάνει. Τι εννοώ. Την αφήνουμε να κάνει οικονομική πολιτική, αλλά όχι πολιτιστική πολιτική. Δεν την αφήνουμε. Δεν της το επιτρέπουμε. Ξέρω ότι η συζήτηση δεν είναι απλή εδώ. Εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε πολιτιστική πολιτική, κοιτάξτε τα πνευματικά δικαιώματα ή στη Γερμανία τώρα γίνεται συζήτηση για το ε, θέμα του ΦΠΑ στις οικαστικές τέχνες και μας ε, απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πάει στο δικαστήριο. Ένας χαμηλός φορολογικός ε, συντελεστής έχει σημασία και δεν μπορούμε να πάμε από 7% στο 19%. Ε, αυτό είναι πολιτιστική πολιτική, δεν είναι μόνο οικονομική πολιτική. Αλλά είναι μια πολιτιστική πολιτική που δεν εγγράφεται ε, υπό την επικεφαλίδα, ούτε ε, θεωρείται ως τέτοια, ούτε συζητείται καν. και στη Γερμανία το συζητούμε στις πολιτιστικές ενώσεις. Και λέμε ότι δεν επιτρέπεται να γίνει κοινοτική και η αρχή της επικορικότητας είναι πραγματικά εδώ το αποφασιστικό στοιχείο. Αλλά πιστεύουμε ότι αν προχωρήσουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα προγράμματα που προωθούν τον πολιτισμό, και τον ενισχύουν οικονομικά, θα πρέπει σε κάποιους τομείς να βάζουμε ε, το κέντρο βάρου στον πολιτισμό και να επιτρέπουμε πολιτιστικές συζητήσεις. Γιατί η συζήτηση για το νέο πρόγραμμα για την ε, δημιουργική Ευρώπη θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει και αυτή η συζήτηση. Το θεωρούμε <coughs> ως μεγάλη ευκαιρία να αυξηθεί και η περικοδότηση 37% αύξηση είναι πολλά λεφτά και το υποστηρίζουμε. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα το βρίσκαμε θαυμάσιο, υπέροχο, αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι παρόλα αυτά παραμένει πολύ μικρό το πρόγραμμα. Ακόμα και αν μας χαροποιεί τόσο ε, θετική αύξηση. Και στη Γερμανία κυρίες και κύριοι έχουμε μια παροιμία που λέει Κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά μέχρι τώρα το πρόγραμμα από την ίδια την ιδέα του είναι πέντε και στο χέρι. Τώρα μπορεί να μας περισσότερα ε, και μεγαλύτερη πρικοδότηση ε, θα είναι πέντε ακόμα, δεν θα έχουν γίνει δέκα, αλλά θα είναι πιο ωραία αυτά τα πέντε. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στα δέκα αυτή είναι η πολιτική που μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσίμερμαν. Τα δέκα είναι στα χέρια των καθαρών συνεισφορέων, αυτές οι χώρες που πληρώνουν. Το είπαμε. Γερμανία, Ολλανδία. Ποιος άλλος είναι. Και αυτοί δεν είναι πρόθυμοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αφήστε δε που θέλω να κάνουν και περικοπές. Και θα πρέπει ε, να φροντίσουμε αυτό το λιγότερο να μην πλήξει την ε, παιδεία και τον πολιτισμό. Εκεί ε, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε μαζί και ελπίζω να μας βοηθήσουν και η Δανική Προεδρία και η επόμενη από αυτό το κουρβανά, το πορτοφολάκι βασικά, να βρούμε τα χρήματα. Εγώ ξέρω που θα τα έκοβα, αλλά δεν το λέω τώρα εδώ. Ευχαριστώ κύριε Τσίμερμαν και έρχομαι στον καθηγητή κύριο Ντέιβιτ Χες επικεφαλής του Ινστιτούτου ε, ε, Επιστημών Κοινωνίας και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λίτς. Έχετε το λόγο. Μα τι τίτλος είναι αυτός για ένα τόσο νέο άνθρωπο, τόσο μακροσκελής. Let me start by saying... Ευχαριστώ να πω ότι το πρόγραμμα για τη δημιουργική Ευρώπη δικαιολογείται γιατί θα πρέπει να δούμε και τους μη ε, και τη μη διάσταση, αλλά και την δυνατότητα, την εμπορική τη ψυχαγωγία και τη δημιουργία στην Ευρώπη σε ένα κοινό πλαίσιο. Και οι δύο τομεί έχουν να κάνουν με την παραγωγή άειλων αγαθών και την κάλυψη πνευματικών αναγκών. Συνδέονται με το γεγονό ότι ανταγωνίζονται για το ίδιο μερίδιο αγορά ελεύθερου χρόνου των πολιτών. Και βεβαίω και δαπανών βεβαίως επικριτικά σχόλια για το τρέχον πρόγραμμα. Ε, σωστά είναι, διότι ασχολούνται και με το καθεστώς των ανισοτήτων των ευκαιριών που μπορεί να παρέχονται από τη μια για τον πολιτιστικό τομέα και για τον εμπορικό δημιουργικό τομέα από την άλλη. Εφόσον καθορίσουμε τις λεπτομέρειες για το μελλοντικό πρόγραμμα του δημιουργικού τομέα και του ακουστικού θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια ζητήματα. Οι προτάσει για την δημιουργική Ευρώπη απηχούν πολλέ από τι πρόσφατε εξελίξει τη ε, πολιτικέ παγκοσμίω και το τι γίνεται με το δημιουργικό κλάδο. Έτσι λοιπόν το ιστορικό και οικονομικό πλαίσιο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εγώ προτιμώ τον όρο πολιτιστικό κλάδος και αυτόν θέλω και να χρησιμοποιήσω σήμερα. Το αποτέλεσμα της αύξησης του ελεύθερου χρόνου και της εξάπλωσης των τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει στην ε, έκρηξη των ε, πολιτιστικών βιομηχανιών και των κλάδων τους τον, τελευταίο, τον προηγούμενο μάλλον αιώνα. Έτσι λοιπόν ανθίζουν οι κλάδοι αυτοί, αλλά υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση, συνάθρηση και κάθετη ομαδοποίηση σε όλους τους τομείς του κλάδου. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Αλλά το τομέας της ψυχαγωγίας είναι επιρρεπής σε αυτή την τάση. Διότι υπάρχει υψηλό κίνδυνος στον κλάδο αυτό. Ακριβώς γιατί η ζήτηση είναι τελείως απρόβλεπτη για τα πολιτιστικά αγαθά. Όπως είπε και ο Βίλιαμ Γκόλντμαν κάποτε, για το λόγο που είναι πετυχημένα σε κάποιες ταινίες και κάποιες όχι, απάντησε κανείς δεν ξέρει. Πρόσφατα, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι τάσεις συγκέντρωσης έχουν λάβει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στο χώρο. Οποιοςδήποτε, οπουδήποτε, μπορεί να γράψει μουσική ή να συγγράψει ένα αφήγημα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει αποκέντρωση τον κλάδο αυτό. Όμως, αντιθέτως, υπάρχει σοβαρή συγκέντρωση των πόρων και των επιρροών. Νέα Υόρκη και Λονδίνο για τη μουσική, Χόλιγουντ για τον κινηματογράφο και το καθεξής. Ακόμα και οι εξελίξεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διάφορες περιφέρειες καθορίζουν τις ανάγκες, τις νέες ανάγκες της ε, ε, πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιστορικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά οι κυβερνήσεις έχουν επιδοτήσει τις τέχνες που χρειάζονται στήριξη, ώστε να προωθηθεί η εθνική ταυτότητα και η ευημερία των πολιτών. Κάποιες φορές βέβαια αυτό φαίνεται ότι φαινόταν να, τα πολιτιστικά αγαθά φαινόταν να είναι προνόμιο των λίγων. Στα τέλη του 20ου αιώνα η παραδοσιακή πολιτιστική βάση βεβαίως έχει παρακμάσει και υπήρξαν και λαϊκιστικές επιθέσει επιθέσεις στον ε, πολιτιστικό χώρο. Ζήτησαν λοιπόν κάποιοι επιδοτήσεις της τέχνης να εγκαταλειφθούν, διότι η πολιτιστική παραγωγή μπορούσε να αυτό τροφοδοτηθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο. Εδώ η πολιτιστική πολιτική άρχισε να αλλάζει στον ε, πολυπολιτισμικό κόσμο. Διότι ο νεοφελευθερισμός και τα υπόλοιπα στοιχεία του σύγχρονου κόσμου βασίζουν την ε, στήριξη της τέχνης σε οικονομικά επιχειρήματα. Εδώ ο στόχος της πολιτιστικής ε, πολιτικής πολλές φορές πρέπει να καλύψει την απέτηση δημιουργίας θέσεων εργασίας όπως ε, συμβαίνει ακριβώς σήμερα με τον τομέα της δημιουργίας και της ψαγωγίας στα τέλη του 20ου αιώνα, την δεκαετία του 90. Πόσο ακριβείς λοιπόν είναι τέτοιες τοποθετήσεις για τον έμεσο και άμεσο αντίκτυπο της τέχνης την ε, στον κλάδο της δημιουργίας. Οι διάφοροι δείκτες, οι μετρήσεις, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η, ο ρυθμός της ανάπτυξης ε, κάποιες φορές έχει υπερεκτιμηθεί. Όμως, σε περιοχές όπως η Ευρώπη, ο τομέας της δημιουργίας εξαπλώνεται σταθερά, τουλάχιστον σε σχέση με του υπόλοιπου τομεί τη οικονομία. Και αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική, ενιαία πολιτική για, την, για τον κλάδο τη δημιουργία. Όχι μόνο για να εντοπίσουμε και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά να καλύψουμε και τις εξελίξεις και την ανάπτυξη που ζητά αυτός ο γοργά εξελισσόμενος τομέας. Η Ευρώπη έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου ω προ την καλλιτεχνική και δημιουργική παραγωγή λόγω τη υψηλή εκπαίδευση, ε, τη ε, διατήρηση τη ε, πολιτιστική κληρονομιά και των αστικών κέντρων όπου υπάρχει σαφής καλλιτεχνική παραγωγή. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει μια τέτοια πολιτική για να δημιουργήσει και άλλες θέσεις εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του 2020. Ωστόσο, και εδώ θέλω να περάσω στο δεύτερο μέρος της ε, παρουσίασής μου, το πώς θα ορίσουμε τις επιδοτήσεις για τον πολιτισμό βάσει μόνον οικονομικών στόχων, αυτό μπορεί να βλάψει τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρουν τέχνη και ο πολιτισμός. Την ανθρώπινη δηλαδή ανέλυξη και το πόσο μπορούν τέτοια ωφέλη να διατηρηθούν εντός εμπορικού συστήματος. Υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στις σύγχρονες κοινωνίε που δεν επιτρέπουν στον πολιτισμό και τις τέχνες να συμβάλλουν στην ανθρώπινη, στην εξέλιξη του ατόμου. Πρώτα απ' όλα οι ανισότητες από την πλευρά της ζήτησης η πρόσβαση του κοινού και η συμμετοχή καθώς και ο αποκλεισμό από τον πολιτισμό είναι ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό. Οι σχεδιαστές πολιτικών έχουν πιέσει τα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα με απαραίτητη χρηματοδότηση και προσπαθούν να καλύψουν όλο το δυνατόν και ε, περισσότερο μέρο του κοινού η πολιτιστική πολιτική πάντοτε πρέπει να συνδυάζεται και με άλλου πολιτικού τομεί, ιδίω την εκπαίδευση, προκειμένου να, καταπολεμά, να καταπολεμάται ο αποκλεισμό και να καλύπτονται οι ανάγκε των ε, ομάδων με μειονεκτήματα. Η κλάδε τη δημιουργία μπορεί να χρησιμοποιούν μεθόδου τη αγορά για νέα μερίδια τη αγορά ή του κοινού και αυτό φαινομενικά φαίνεται να λειτουργεί, αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Διότι δεν λειτουργούν τα άλλα αγαθά όπως τα κλασικά εμπορεύματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θέλουμε να καταρτήσουμε με την πολιτιστική πολιτική για την Ευρώπη. Επίσης υπάρχει ανισότητα και στην πλευρά της προσφοράς. Υπάρχει αυτό το στοιχείο που ανέφερα και προηγουμένως, υψηλός κίνδυνος στον τομέα της ψυχαγωγίας και της δημιουργίας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σαφείς τάσεις ε, συγκέντρωσης στην αγορά και στο χώρο. Στις ε, μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί τελικά εφόσον υπάρξει σωστή στήριξη να αναλογεί και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και του κοινού. Εδώ θα μπορούσε λοιπόν ο κλάδος της δημιουργίας να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντική άνθηση. Εδώ τώρα θα ήθελα να αναφέρω και μερικά προβλήματα υλοποίησης. Τα μέσα επικοινωνίας θα πρέπει να μας βοηθήσουν να αποκοινούμε τα ψυχαγωγικά μας μέσα να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα κενό, κενά. Εδώ μπορεί να υπάρχουν και πολιτιστικές διαφορές βέβαια που θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό για να βεβαιωθούμε ότι το δυναμικό του τομέα της δημιουργίας αξιοποιείται και το εξειδικευμένο προσωπικό αυτού του κλάδου να καλύψει και τις μη κερδοσκοπικέ ανάγκες του τομέα. Τέλος, να επιστρέψω στα προβλήματα των αγορών στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δεν έχω τοποθέτηση κατά της αγοράς εξ αρχής εδώ. Αναγνωρίζουμε ότι πολλές φορές η αγορά μπορεί από μόνη τη να οδηγήσει στην παραγωγή εμπορευμάτων και αγαθών που βελτιώνουν την ευημερία των ανθρώπων. Αλλά κάποιε φορέ αυτό δεν πετυχαίνει. Οι οικονομολόγοι και οι κοινωνιολόγοι έχουν αποδείξει ότι πολλά χαρακτηριστικά των κλασικών αγορών καθιστούν τους μηχανισμούς της αγοράς ακατάλληλους για την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως οι Beatles ή ο Μανού Τσάο. Εδώ δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών. Υπάρχει τάση των πολιτιστικών αγαθών λειτουργούν ως δημόσια αγαθά και υπάρχει και υψηλό ποσοστό σταθεροποίησης του περιφερειακού κόστους. Τα βαθύτερα προβλήματα και αίτια της αποτυχίας της αγοράς των τομέα των πολιτιστικών ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι ζωτική σημασία οι επιδοτήσει των κυβερνήσεων, οι κρατικέ επιδοτήσει. Δύο τελευταίε παρατηρήσει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, ο κλάδο τη δημιουργία μπορεί να αυξάνεται σταθερά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σε αυτό τον εξελισσόμενο τομέα με υψηλό κίνδυνο κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και μάλιστα βιώσιμε. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής σε αυτόν τον κλάδο δεν είναι υψηλή. Όπως ας πούμε ο ανεξάρτητος ε, τομέας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι πολύ επισφαλής η θέση εργασία σε ένα τέτοιο κλάδο. Σε ποιον λοιπόν βαθμό η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και της ψυχολογίας θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με το πρόβλημα των εγγύσεων. Διότι πολλές φορές οι τάσεις μόκλευσης δεν αποδεικνύονται. Επίσης υπάρχει και ένας ολόκληρος χώρος μεσαζόντων που τελικά δεν ανήκουν στο χώρο του πολιτισμού. Καθώ αναπτύσσεται ο επόμενο κύκλο ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές για να πάυσουν οι άστοχες κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά λοιπόν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο πολιτισμός να καλύπτονται από το ίδιο πρόγραμμα μπορεί από πολλές απόψεις να είναι ευπρόσδεκτα. Όμως το Κοινοβούλιο ας κάνει ό,τι μπορεί ώστε ο μη κυρδοσκοπικός και έξω θεσμικό τομέας θα προστατευτεί από τις δυνάμεις της αγοράς και ότι θα διατηρηθεί το μεγάλο δυναμικό του κλάδου της δημιουργίας. Very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Πάρα πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε και ορισμένα από αυτά που είπατε στο τέλος είναι ακριβώς και δικά μας μελήματα, βασικά. Θέλουμε να δουλεύουμε σε μικρότερη κλίμακα αλλά έχουμε το πρόβλημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δουλεύει σε μεγάλη κλίμακα, χονδρικά, για να μην έχει πάρα πολλά μικρά ποσά και να ελέγχει πού πηγαίνουν. Εμείς προτιμούμε 200.000 300.000 αντί 20 10 ε, ή λιγότερο. Αυτό προτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 200 και 300 Αυτό είναι το πρόβλημα στον πολιτισμό. Τα μεγάλα ταμεία, τα περιφερειακά έχουν τεράστια ποσά και είναι και πιο εύκολο για τους υπαλλήλους να τα κοιτάνε και να τα χειρίζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στον κύριο Ράντου Μαχαηλιανού, το σκηνοθέτη μας και επίτιμο πρόεδρό μας της ε, Επιτροπής ε, του βραβείου Λουξ. Παρακαλώ. Ε, bonjour. D'abord un grand grand merci de nous accueillir. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας υποδέχεστε και μας Ούτε εγώ είμαι σκηνοθέτης, ε, γράφω σενάρια, είμαι και παραγωγός. Και αν ε, συνεργαζόμαστε εδώ και καιρό είναι γιατί βασιζόμαστε σε εσά για να αλλάξουμε το ρεύμα και αν ακόμη είμαστε μερικές φορές ε, απεσιόδοξοι σε αυτές τις σκληρές εποχές πρέπει να κρατήσουμε ένα πνεύμα αισιοδοξία. οι συνάδελφοι μίλησαν πολύ για τεχνικά ζητήματα. Εγώ θα κοιτάξω να πω άλλα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά θα θυμίσω μερικά νούμερα. Όλοι ξέρουμε ότι ο κόσμος και η Ευρώπη περνάνε μια πολύ δύσκολη στιγμή οικονομικής κρίσης. Οπότε άμα το δει κανείς απ' έξω και από μακριά φαίνεται παλαβό να, να, να, να ζητήσει κανείς μια αύξηση και να την πάρει όταν όλοι σφίγγουν το ζωνάρι. Να θυμίσω όμως έναν αριθμό. Η πρόταση για τον προπολογισμό για τον πολιτισμό είναι το 0,02% του συνολικού προϋπολογισμού. Όταν ο τομέας του πολιτισμού είναι πάνω κάτω το 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και, και απασχολεί το 3,8 των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 8 και κάτι εκατομμύρια κόσμο. Και αναρωτιέμαι, ποιες είναι οι προκλήσεις, δεν είναι τεχνική ερώτηση, ποιες είναι οι προκλήσεις για μας πολίτες της Ευρώπης ε, και μας τους καλλιτέχνες ε, που είμαστε πρωταγωνιστές ε, του πολιτισμού και της ε, πολιτικής για να δράξουμε αυτές τις ευκαιρίες. Αυτός ο κόσμος είναι πραγματικά ε, παθιασμένος, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πάρα πολύ μπερδεμένο. και ο ρόλος μας είναι να διαδώσουμε τον πολιτισμό ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να καταλάβουν την πολυπλοκότητα της, κατα της κατάστασης και να μπορούν να ζήσουν σε αυτόν τον ε, πολύπλοκο κόσμο. Είναι πρωταρχικό πράγμα ο πολιτισμός, γιατί μέσα από τη γνώση, την ευφία και τον πολιτισμό θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για όλα τα υπόλοιπα. Και μέσα από τον πολιτισμό επίσης θα δημιουργήσουμε κοινωνικούς δεσμούς όταν ο κόσμος ε, ε, σε πολλούς ε, τομείς αρχίζει και κλείνεται και σφίγγεται. Τις προάλλες ρώταγα του μπαμπά μου, ο οποίος είναι κοντά στα 91 και ο οποίος έχει διασχίσει όλη την Ευρώπη. Εμείς είμαστε μεν Ρουμάνοι, αλλά ο μπαμπάς μου έζησε το φασισμό, τον πόλεμο, τον σταλινισμό, τον Τσαουσέσκου, τη δικτατορία του και εδώ και 20 χρόνια έχει την τύχη να ζει στη Γαλλία και τον ρώτησα έτσι ανησυχώντας ε, με όλα αυτά που μας ανησυχούν όλους τον ερώτησα ο κόσμος στα νιάτα σου ήταν πιο βίαιος από ότι ο κόσμος σήμερα ο κόσμος στα νιάτα σου ήταν πιο ευφύης από ότι ο κόσμος σήμερα και μου απάντησε και μ' άφησε έκπληκτο ότι ο κόσμος στα νιάτα του ήταν πολύ πιο βίαιος. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα ήμασταν ε, πιο βίαιοι. Μου είπε ότι η Ευρώπη ήταν συνέχεια επιποδός πολέμου με τεράστιες κοινωνικές αντιμαχίες και μου είπε ο κόσμος σήμερα είναι πολύ πιο έξυπνος, πιο ευφύης ε, τεχνολογικά και επιστημονικά αλλά είναι πολύ λιγότερο ευφύης δυστυχώς στο πνευματικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Και εδώ πάλι αναρωτήθηκα κάτι. Τι είναι το πνευματικό, μιλάμε για το κοσμικό πνευματικό, δεν μιλάμε για το θρησκευτικό πνευματικό σκέλος. Και αναρωτήθηκα εκεί όπου πραγματικά έχουμε ελλείμματα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στο κοσμικό ε, πνευματικό ε, τομέα, είναι ο ρόλος του πολιτισμού να μπορέσει να εξάρει τους ε, ανθρώπους και να τους ε, ε, φέρει στο διάλογο με το άπειρο, ε, όχι δηλαδή να τους βγάλει από το πεπερασμένο και από τη σχέση με το κορμί τους και με το μικροχώρο τους. Δηλαδή δεν έχουμε την αντίδραση που μπορεί να, να παλέψει με τον ηλισμό και τον φονταμενταλισμό που ε, αντιπαλεύουν ακριβώς αυτό το ε, κοσμικό πνευματικό στοιχείο. Η ποιότητα λοιπόν της γνώσης, η ποιότητα του προβληματισμού και της σκέψης είναι η πρόκλησή μας. Η πρόκληση για να βγούμε από την κρίση και να βοηθήσουμε τον κόσμο είναι να αυξήσουμε ε, την, ε, τον προϋπολογισμό στον πολιτισμό και για τη δική μας τη γενιά και για τις μελλοντικές γενιές. Και όπως υπόθηκε σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που έχουμε σήμερα, Ευρώπη και Αμερική από τη μια και Ασία από την άλλη, εμείς είμαστε η παγκόσμια αρχηγοί ακόμα. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον τομέα για να κυνηγήσουμε άλλους ε, τους οποίους δεν θα ξεπεράσουμε πολλές φορές όπως με στην τεχνολογία για ορισμένες παραγωγές. Ενώ στην κουλτούρα, στον πολιτισμό είμαστε πάντοτε αρχηγοί. Και αυτό το οποίο είναι μια τρομερή τύχη για μας και ένας απίστευτος πλούτος είναι η πολυμορφία, ο πλούτος της Ευρώπης και η ιστορία της. Λοιπόν, και τώρα για να ξαναπροσγειωθώ ε, έναντι της πρότασης της Κομισιόν όπως και οι συνάδελφοι υποστηρίζω πάρα πάρα πολύ. Εδώ και μισή χρόνο συζητάμε και με την Επίτροπο για τον Πολιτισμό και, για τον και με τον κύριο Μπαρόσο. Είναι η ανεξαρτησία του προγράμματος Μέντια και ως προς την αποστολή του και ως προς τον προϋπολογισμό του. Και όχι μόνο να είναι ανεξάρτητο το Μέντια, αλλά και στο εσωτερικό του να έχει καθαρά και εξάστερα την υποδιέρεση των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού, κατανομή, παραγωγή και, διανομή, παραγωγή κτλ. Και αυτό δεν το λέω από εγωισμό, γιατί το, με αίσθημα δικαιοσύνη το λέω. Διότι σήμερα τα οπτικακουστικά μέσα και ο κινηματογράφος είναι ο μεγαλύτερος ε, παιδαγωγικός φορέας στην Ευρώπη. Όταν ε, εμείς αρχίζουμε και ανακατεύουμε εδώ όργανα και άτομα ε, βρισκόμαστε σε πλήρη ψηφιακό αναβρασμό. Τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε κάτι, τρέχουμε από πίσω γιατί δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά τι γίνεται. Λοιπόν, είναι όλα αυτά πάρα πολύ ιδιόμορφα. Το να συζητάει κανείς με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε με ανθρώπους από το θέατρο, την όπερα ή τη μουσική, για κάτι τόσο το συγκεκριμένο σε πλήρη ε, επανάσταση, ε, αυτό θα ήταν ένα πραγματικό λάθος. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο λειτουργήσε από το 2007 και μετά πάρα πολύ καλά, την αξερτησία του προγράμματος και, την, και τον του προπολογισμού του και όπως επίσης και τις υποδιαιρέσεις μέσα στον προπολογισμό. Και να σας αναφέρω και ένα τσιτάτο του Βικτόρ Ιγκό που στην, το 1848 στις 10 Νοεμβρίου στη Εθνοσυνέλευση. Ήδη ψήφισα και θα συνεχίσω να ψηφίζω όλες τις περικοπές που προτείνονται, εκτός από εκείνοι που αποτελούν την πηγή του δημόσιου βίου. Και λέω κύριοι ότι οι μειώσεις στον προϋπολογισμό για τις επιστήμες, τα γράμματα και την τέχνη είναι καταστρεπτικές θα, σε, από όλες τους τις πλευρές. Τι θεωρείτε εσείς κύριοι για κάποιον έναν ιδιώτη που έχει 1500 φράγκα εισόδημα και θα διέθετε από την περιουσία του μόνο 5 φράγκα το χρόνο για την παιδεία και θα ήθελε όταν κάνει οικονομίες να εξοικονομήσει δραχμοδί φράγκα πάνω στην ευθεία του την ίδια. Ποιος είναι ο κίνδυνος σήμερα Σήμερα ο κίνδυνος είναι η αμάθεια. Η αμάθεια είναι μεγαλύτερος κίνδυνος, μεγαλύτερος και από την μιζέρια. Η αμάθεια που μας κατακλίζει και μας πολιορκεί από παντού διότι μέσω της αμάθειας περνάνε παράλογες θεωρίες ε, στα κεφάλια των ανθρώπων και σε μία τέτοια φάση σε μία τέτοια στιγμή τολμάμε εμείς ε, να ευνουχίσουμε όλα αυτά τα θεσμικά όργανα τα οποία έχουν ως στόχο την καταστροφή της αμάθειας. Ε, Merci Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσουμε πολύτιμα αυτά τα λόγια του Βίκτορο Σουγκό, που θα μπορούσαμε να τα γράψουμε λίγο πιο σύντομα και θα τα διαβάσουμε στους υπουργού οικονομικών και στους καγκελαρίους, στις καγκελαρίους, πώς τους λένε εκεί τους κυβερνώντες. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε γιατί ε, είστε και επίτιμος πρόεδρος της κριτικής μας επιτροπής για το βραβείο Λουξ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες υπόθηκαν τα περισσότερα. Στι συζητήσει θα μπούμε σε επιμέρους λεπτομέρειε. Παρακαλώ, συνάδελφοι, τώρα να μην επαναλάβετε όλοι τα πάντα, γιατί θα τα συζητήσουμε ξανά τα θέματα αυτά. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κώστα μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι κάτι το διαφορετικό από εμπειρογνώμονες. Είναι άνθρωποι του πολιτισμού, είναι άνθρωποι με μεγάλο περιεχόμενο και βάθος. Είμαι συγκινημένη από αυτά τα οποία άκουσα τελευταία από τον Ράντου Μιχαλιάνου. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μία τεράστια πρόκληση μπροστά μας. Την πρόκληση του οικοδομήσουμε έναν ορίζοντα για έναν, για έναν ναι, ουμανισμό που θα συμμερίζονται όλοι άσχετα από το αν θα είναι λαϊκοσμικός ή όχι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να, γίνει, να γίνεται όλο ένα και πιο κεντρικό στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Ξεκινώντας από ένα θετικό στοιχείο Πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι έχοντας βέβαια και τη συνέστηση των προκλήσεών μας απάντη, μπροστά μας. Έχουμε έναν ορίζοντα μεταρρυθμίσεων που ακόμη και οι χρήστες προσπαθούν να ερμηνεύουν πάνω στη βράση ενώ εργάζονται και Θεωρώ ότι η πράσινη βίβλος ε, για τους οικονομικούς κλάδους δημιουργίας, ε, ε, για την κουλτούρα, στενή τη έννοια και για την τεχνολογία προσπαθούν να τεντάξουν όλα αυτά. Εδώ μιλήσαμε ότι με αυτήν την πρόταση είμαστε στο 0, Πέντε, δεν έχουμε βέβαια μηδέν ακόμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο μηδέν μπροστά μετά το κόμμα, συγγνώμη. Ελπίζουμε όμως οι ελπίδες μας να μην καταστραφούν, ελπίζουμε οι υπουργοί να μην μας διαψεύσουν. και ο νέος προγραμματισμός ε, της Κομισιόν αυξάνει κατά 7% και τα κονδύλια για τον πολιτισμό και για την εκπαίδευση και την παιδεία. Τώρα τρία-τέσσερα σημεία. Λοιπόν, έλεγα, συμμερίζομαι τις ε, απόψεις ε, του κυρίου Ζήμερμαν σχετικά με την τοποθέτηση αυτού του προγράμματος. Η εξαφάνιση του, από τον τίτλο της λέξης ε, «κουλτούρα» μπορώ να το καταλάβω γιατί θέλει να, να δώσει έναν τίτλο πιο σύντομο αλλά δεν θα ήθελα ο πολιτισμός, η κουλτούρα να μπει στο περιθώριο. Και σε αυτό το πρόγραμμα η αξιοποίηση των πολιτιστικών διαφορών και του διαπολιτιστικού διαλόγου δεν είναι τα μόνα στοιχεία. Αλλά ε, θέλουμε να μην έχουμε μια οικονομιστική προσέγγιση της κουλτούρας, αλλά να ενισχύσουμε και την αμοιβαία ε, αξία ε, του πολιτισμού και να δημιουργήσουμε συνέργεια μεταξύ του ευρωπαϊκού πολιτισμού υλικού και αϊλού. Μια άλλη διάσταση που κάποιος από εσά την ανέφερε και που συμμερίζομαι είναι η διάσταση local που αναφέρατε, η διάσταση, η τοπική διάσταση και η εμπλοκή της, ε, των κλάδων οικονομικής ε, δημιουργίας ε. με την εμπλοκή των, του, τοπικού δυναμικού της Ευρώπης, χωρίς όμως να πέφτει στον τοπικισμό. Έχουμε μία ευρωπαϊκή πρόκληση. Και έτσι λοιπόν και για την ψηφιοποίηση των αιθουσών από τη μια και το θέμα της εναρμόνισης του ΦΠΑ για τα πολιτιστικά προϊόντα, τις εκδόσεις κτλ. Όλα αυτά θα μπορούσε να, επιταχυνθούν. Το merging του ολοκληρωμένου προγράμματος της Κομισιόν. Καταλαβαίνω ορισμένες απαιτήσει. δεν θα μακρηγορήσω αλλά δράτω με μεγάλη προσοχή και το συζητήσαμε και με τους συναδέλφους, το γεγονός ότι για να μειώνοντας τα δύο προγράμματα πολιτισμό και ε, οικονομικό κλάδο της δημιουργίας και το μέντια να τα ενώσουμε θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας περισσότερο κινδύνου και όχι θετικών αποτελεσμάτων. Εγώ εισηγήτρια είμαι και θα το αναλύσω καλύτερα και θα ήθελα να, αναλύσω, να αναλύσουμε και όλες τις πτυχές όπως είπε και ο σκηνοθέτης προηγουμένως. Για το θέμα του καθηγητή Καρούζο και του καθηγητού από το Λίτς. Το νέο σενάριο προβλέπει μία εγρήγορση των network έναντι των παραγωγικών μορφών παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης. Ερώτηση. Κύριε Καρούζο, αλλά και οι υπόλοιποι, άμα δούμε σήμερα τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε, η Ευρώπη πρέπει να συνοδεύσει αυτή την αλλαγή. Δεν μπορεί να κάνει άλματα στα τυφλά. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια και ενίσχυση των εξαρτήτων παραγωγών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μποχλός σε εθνικό επίπεδο είναι οι δημόσιες και εν μέρει ιδιωτικές τηλεοράσεις που επενδύουν ε, ιδιαίτερα στην κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Ρωτώ. Η δυνατότητα του δικτύου να μην έχει μόνο ένα ρόλο ε, παραγωγής ε, Ε, ε, διανομής συγγνώμη, ε, των διαφόρων έργων που διαδίδονται, ξέρουμε πολύ καλά, και μέσα από πειρατικές μεθόδους σε μεγάλο βαθμό. Και όχι πια τόσο ρόλο, μεγάλο ρόλο στην παραγωγή. Μήπως θα έπρεπε να γίνει και ένα άλμα και να φανταστούμε επενδύσεις ή τουλάχιστον μία ποσόστοση χρηματοδότησης που θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τους ε, ε, ε, χρήστες, ε, για, για τους, συγγνώμη, τους λειτουργούς των δικτύων. Βλέπετε πέφτουν από παντού τα έσοδα, μήπως και από εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποιου, κάποιους πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να μην μακρηγορήσουν. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, παρακαλώ, στους εμπειρογνώμονες, γι' αυτό τους καλέσαμε, για να μας ε, βοηθήσουν να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις μας. Ο κύριος Βέρα από τη Σλοβενία, παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να φύγω για να μην χάσω το αεροπλάνο μου. Για να σας πω σύντομα το εξής. Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι πολύ δαπανηρά σε αυτά τα προγράμματα. Και εμείς πώς μπορούμε να προωθήσουμε την παραγωγή και τη δημιουργία των μικρών δημιουργών. Αυτό που λέμε θετική διάκριση. Να τους βοηθήσουμε ε, για να βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνες τις χώρες που έχουν ε, μια ε, πολύ ε, έντονη δημιουργική παραγωγή. Δίνει τη δυνατότητα το παρόν μέσο ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν και αυτοί μια καλή πρόσβαση στον πολιτισμό, δηλαδή στην ενίσχυση, την οικονομική. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία και με εγγυήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και γεωγραφικά θα πρέπει να γίνει καλή επιλογή των τραπεζών εκείνων που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν καλή πρόσβαση από το Ταμείο αυτό των εγγυήσεων. Οι πιστώσεις στη συνέχεια χορηγούνται από τις εκάστοτε τράπεζες των διαφόρων χωρών ε, ή των γειτονικών. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη, πρέπει οπωσδήποτε να φύγω και δεν θα περιμένω την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Και να ευχαριστήσω και εσένα, Ντόρι, που μα επέτρεψε να ακούσουμε δημοσίω τι απόψει τέτοιων εμπειρογνωμόνων, που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένε και είναι ιδιαίτερη ε, ιδιαίτερα ενδιαφέροντε. Επίση, να πω πόσο θαυμάζω τον σκηνοθέτη μα τον κύριο Μιχαλιάνου και πόσο σημαντικό τον θεωρώ. Να πω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να ενισχυθεί ο τομέα και του πολιτισμού και τη δημιουργία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη ψηφιακή εποχής. Άκουσα τι είπατε για τα χρηματοδοτικά και οικονομικά μέσα που θα πρέπει να αποδοθούν στον τομέα του πολιτισμού. Όμω είναι μεγάλη απογοήτευσή μου διαβάζοντα τι λεπτομέρειε αυτού του προγράμματο και δεν θα την ξεπεράσω εάν τα πράγματα μείνουν ω έχουν. Εδώ κυριαρχεί το πνεύμα τη ανταγωνιστικότητα τη αγορά και στήριξη του τομέα. Αυτό καλό είναι. Όμω δεν βλέπω καμία αναφορά στην αξία του πολιτισμού και την δυνατότητα που έχει ή ε, που μπορεί η δημιουργία να προσφέρει και στην πολιτική συνείδηση και στις ανθρώπινες αξίες. Αυτή θα πρέπει να είναι η πραγματική ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως είπε και ο κύριος ε, Μιχαλεάνου. Τα υπόλοιπα θα είναι σαν ένα καρναβάλι στο οποίο δεν θέλω να συμμετάσχω. Τώρα, ω προ την οικονομική αύξηση, που θα είναι βιώσιμη και χωρί αποκλεισμού, ουδέποτε γίνεται λόγο για κάποιο μοντέλο. Για το κατά πόσον ανήκουμε σε μια κοινωνία πολιτιστική, με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Παρά λοιπόν την θέλησή σα να αξιοποιήσετε στο δυνατόν καλύτερα του πόρου προ όφελο των προγραμμάτων που θα στηρίζονται, εγώ θέλω να ζητήσω να δώσετε προσοχή σε πολλά σημεία τα οποία θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, ο οικονομικό προσανατολισμός που θα δίνεται στα προγράμματα μπορεί να βλάψουν τα πολιτιστικά του ωφέλη, δηλαδή χρηματοδότηση σχεδίων με μεγαλύτερη απόδοση οικονομική και όχι πολιτιστική. Αυτό φαίνεται ότι θα πρετανεύσει στι επιλογέ σα. Έπειτα, οι διατάξει όπω έχουν περιληφθεί στον κανονισμό. Αυτέ είναι τόσο ασαφείς, τόσο πολύ ασαφείς, που πραγματικά δεν προσφέρουν σε κανέναν, σε, σε πραγματικά κανέναν, καμία εγγύηση για το πώς θα εκτελεστεί σωστά το πρόγραμμα. Και εδώ πραγματικά προειδοποιώ επισήμω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα αφήσουμε να περάσει έτσι. Ένα τέτοιο κενό, μια τόση ασάφεια. Επίση, ο κανονισμό δεν δίνει καμία διευκρίνηση για το πώ θα προβλέψει νέο δημοσιονομικό εργαλείο βάσει του διατομεακού ε, κεφαλαίου. Και επίση, σε ποιου πολιτιστικού τομεί θα σταθούμε. Πώ θα καθοριστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πώ θα κατανεμηθούν οι δανειοληπτικέ εγγύσει και ποιο θα έχει την ε, εξουσία για να αποφασίσει ποια θα είναι τα επιλέξιμα προγράμματα και σχέδια. Έπειτα, είναι στεγανά τα δύο τμήματα του πολιτισμού και της, ε, των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αυτό διαφαίνεται από το κείμενο. Ή τουλάχιστον η ασάφεια Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρξει τέτοια, τέτοιος διαχωρισμός. Θα πρέπει επίσης για όσους ανησυχούν για το θέμα αυτό να τους πω ότι χρειάζεται πραγματικά πολύ επιπλέον μελέτη και για τα όσα προβλέπονται για τον προπολογισμό ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι εδώ υπάρχει επαρκή πρικοδότηση. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε καθαρή υποκρισία την οποία θα πρέπει και να αποκαλύψουμε. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, διευκρινίσει ποιο ακριβώς πολιτιστικό εγχείρημα επιδιώκει με το πρόγραμμα αυτά, αυτό. Διότι ούτε με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων και τις παρουσιάσεις τους δεν κατάφερα τελικά να το αποκωδικοποιήσω όλο αυτό. Να με επιτρέψετε πρόεδρε να κλείσω με μια πρόταση. Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι θύμα γενικότερων δυσκολιών, αλλά παραμένω άναυδος και σας παρακαλώ το μεταφέρετε αυτό στην Επίτροπο. Καλό θα ήταν, ήταν και εδώ η ίδια. Λοιπόν, μένω έκπληκτος που δεν έχει προσέλθει. Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε με εκπροσώπου δευτέρα κατηγορία. Θα έπρεπε να είναι εδώ η Επίτροπο. Θα έπρεπε η συζήτηση περί πολιτισμού σε τέτοιε στιγμέ δύσκολη χρηματοδότηση να γίνεται με κάθε σοβαρότητα. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να ξέρει ότι μπορεί να υπολογίζει στη βοήθειά μα, αλλά και εμεί να υπολογίζουμε στη δική τη αφήνεια. Επίση, δημοσίω θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι εδώ έχουμε μια συγκεκαλυμένη περικοπή που επιχειρείται μέσω του προγράμματο πολιτισμού και των ε, μέσων μαζική ενημέρωση. Δεν είμαι αφιλή. Ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει αγώνα εξουσία εντό των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ δύο πόλων που έχουν δημιουργηθεί. Θα ήθελα λοιπόν επισήμω να ζητήσω από την Επίτροπο να, βάλει, ε, να θέσει τέρμα σε αυτέ τι ε, καταστάσει. Διότι ιδάλω θα ζητήσουμε διαφορετικά, θα απευθύνουμε έκκληση στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφορετική χρήση των, και διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων. Και θα πρέπει να πω ότι με την ανάγνωση του κειμένου αυτού δεν βλέπουμε την νομοθετική εγκυρότητα του όλου Η ουσία της δράσης δεν βρίσκεται στις ρυθμίσεις ε, του νομοθετήματος. Ο καθένας στην ουσία θα μπορεί συγκεκαλυμμένα να κάνει αυτό που νομίζει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επικοινωνιακή και μόνο κίνηση εντυπωσιασμό. Αλλά είναι πολύ δύσκολη σε στιγμή για κάτι τέτοιο. Και για να το αφήσουμε να περάσει έτσι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Καβατά. Πολύ βαριά αυτά που είπατε. Όχι ρεαλιστικά, λέει ο κύριο Καβατά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, ε, με γνωρίζετε. Αλλά ε, συμφωνώ μαζί σα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι το κονδύλι. Συζητούμε για ένα ποσό άγνωστο και ποια κονδύλια προβλέπονται για ποιο σκοπό. Και γι' αυτό θέλουμε να εγγραφεί σωστά στον προϋπολογισμό κάθε κονδύλι. Πόσο, για, για ποιο σκοπό, σε ποσοστό. Τώρα δεν έχουμε ποσά. Τα ποσά θα έρθουν αργότερα. Δεν καλέσαμε την κυρία Βασιλείου, γιατί σήμερα κάναμε ακρόση εμπειρογνωμόνων και οι κυρίε και κύριοι που είναι παρόντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνοι που χειρίζονται το πρόγραμμα που το έχουν εκπονήσει και είμαι βέβαιη ότι δεν το έχει κάνει η κυρία Βασιλείου, δεν είναι και δουλειά τη άλλωστε. Βέβαια, εκείνη θα πρέπει να το υπερασπιστεί, έχει δίκιο και να ε, την καλέσουμε στη συνέχεια. Μέχρι το φθινόπερο θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Σήμερα δεν την καλέσαμε. Έχουμε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αυτοί κρατάνε τα ε, στυλό και τα γράφουν αυτά. Ε, η κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβαλε μία αξίωση με το νέο πρόγραμμα για τη βιομηχανία της δημιουργίας και τη δημιουργική Ευρώπη. Θέλει να συνεχίσει και το τμήμα του πολιτισμού, αλλά και στη στρατηγική του 2020 να εξασφαλίσει την ε, ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της δημιουργίας και να την αυξήσει. Για να δούμε όμως αν αυτή η αξίωση είναι πραγματικότητα. Εγώ ισχυρίζομαι πρώτον ότι η πρόταση έχει οδηγήσει σε τόσες συζητήσεις, όχι επειδή ο κλάδος είναι αφελής ή ε, αμαθής ε, ή ε, κυριαρχείται από άγνοια, αλλά είναι τεράστια ασάφεια. Και σας ευχαριστώ όπου δεν απορρίπτεται από χέρι την ε, συγχώνευση των δύο. Αλλά τι γίνεται με ε, το μη εμπορικό κλάδο και με τον εμπορικό κλάδο της δημιουργίας και πώς ε, προστατεύονται αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ο μη εμπορικός κλάδος, γιατί αν δεν προστατεύεται τότε από πλευράς πολιτιστικής πολιτικής δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε τη σημασία της βιομηχανίας και του πολιτισμού και η πολιτιστική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται και θέλουμε να ενισχυθεί βεβαίως, αλλά όχι εις βάρος του βασικού προγράμματος για τον πολιτισμό. Αυτό θα πρέπει να είναι το σαφές μας μήνυμα όταν συζητούμε το νέο πρόγραμμα και πάμε στην επόμενη περίοδο, θυμίζω, ε, τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής ε, ε, ποικιλομορφίας και κληρονομιάς Μπορεί ο πολιτισμός να είναι και εμπόρευμα ε, καμιά φορά, αλλά ε, εκτός αυτού είναι πολύ περισσότερα από εμπόρευμα. Αυτό που είπατε είναι η συνάντηση, η ανταλλαγή, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών, όλα αυτά ισχύουν. Και θα πρέπει να φτάνουμε και σε ανθρώπους και να τους ε, υποκινούμε και να τους παροτρύνουμε να ασχολούνται με το πολιτισμό. Αυτό που ονομάζεται audience building, να δημιουργούμε ένα κοινό για τη δημιουργία αυτή και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο πρόγραμμα και ότι το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πουλάμε ως εμπόρευμα, αλλά ε, πώς θα συμμετέχει ο κόσμος στον πολιτισμό. Να κάνω τώρα την εξής αποφασιστική ερώτηση. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι είναι θέμα ερεσιμότητας, ο μη εμπορικός τομέας ε, του πολιτισμού θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Ωραία. Και μικρά έργα να συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται και όχι μόνο στην οικονομία. Η κυρία Βασιλείου είπε ότι θέλει να βγει επιθετικά, να δώσει περισσότερα χρήματα και όλοι το υποστηρίζουμε και θα ήταν ιδιαίτερα χαρμόσυνο και θετικό αν το καταφέρναμε. Αλλά Έχουμε την κατάσταση στο Συμβούλιο. Οι 8 χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς στην επόμενη περίοδο θέλουν να κάνουν περικοπές 10% στις δημοσιονομικές προοπτικές. Και θέλω να ρωτήσω ειδικά τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν το καταφέρουν αυτό, κινδυνεύει ο προπολογισμό για το πρόγραμμα του πολιτισμού να μην αυξηθεί όπως θέλει η κυρία Βασιλείου και εμείς οι ίδιοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ελπίζω να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Για την περίπτωση λοιπόν που θα γίνει αυτό τι σημαίνει ενδεχόμενη περικοπή, πώς θα επηρεαστεί το πρόγραμμα στην κατανομή των κονδυλίων ανάμεσα στον πολιτισμό, τον αμυγή και τη βιομηχανία της δημιουργίας. Εάν παρελπίδα συμβεί αυτό, πώς θα φροντίσουμε να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα του πολιτισμού. Εγώ θέλω εδώ μια σαφή πολιτική απάντηση, αλλιώς δεν μπορώ να αξιολογήσω πολιτικά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Συμφωνούμε όλοι και προσυγγράφουμε. Πολύ ωραία τα είπατε. Ο Μάρκο Κουρία. <clears throat> Σήμερα θα γυρίσω σπίτι μου ευχαριστημένο. Πρέπει να ευχαριστήσω του τέσσερι εμπειρογνώμονε, γιατί θα γυρίσω πιο πλούσιο στο σπίτι μου. Πιο, πιο πλούσιος σε περιεχόμενα ακούγοντας αυτές τις βαθιές τοποθετήσεις σήμερα το πρωί. Ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι για το πρόγραμμα για τον πολιτισμό και για τα μέντια θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη συμμετοχή των, των no profit, των μη κερδοσκοπικών ε, παραγόνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τους υπόλοιπους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει κίνδυνο στην πρόταση της Κομισιόν να μην διαφυλάξουμε αυτόν τον τομέα. Άλλη μια συνάδελφος, η Πέτρα Καμαέβερτ από τη Γερμανία. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τόσο είπαν οι Συμφωνώ και με τις ερωτήσεις και με όλα. Έχω άλλη μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τους εμπειρογνώμονές μας. Για τη συνένωση των εθνικών οργανισμών. Γιατί ακούμε και εδώ κριτική και μπορώ να την καταλάβω το, για το Media Desk και τα σημεία επαφής για το πολιτισμό αν συγχωνευτούν στον ίδιο φορέα, μα καλύπτουν τελείως διαφορετικούς τομείς. Και θα πρέπει οι ίδιοι άνθρωποι να τα χειρίζονται και υποτίθεται θα οδηγήσει σε συνέργεια και θα βοηθήσει. Δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ. Γιατί ένα μικρό πολιτιστικό πρόγραμμα θέλει άλλη παροχή συμβουλών και συνοδεία και βοήθεια από ότι ένα μεγάλο οπτικοακουστικό πρόγραμμα. Ε, εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Είναι φύση ιδέα πραγματικά να συγχωνευτούν αυτά τα δύο και αν γίνει συγχώνευση ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν και να τους ορίσουμε εμείς έτσι ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά στο μέλλον υπέρ εκείνων που κάνουν τις αιτήσει για να χρηματοδοτηθούν. Ιδιαίτερα υπό το κίνδυνο ότι μικρά πολιτιστικά προγράμματα μπορεί να χαθούν τελείω. Ή, ή οφείλουν ή είναι και πρόθεσή τους, ξέρω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν αλλάζω τη σειρά. Πρέπει να ακούσουμε πρώτα ε, τα δύο άλλα όργανα και μετά τους συμπειρογνώμους. Καλύτερο δεν θα ήτανε. Μάλιστα. Ο κύριος Κρίστενσεν παρακαλώ, εξ ονόματος της Δανικής <coughs> Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω την ε, μετρική μου γλώσσα, εφόσον έχω τη δυνατότητα, να ευχαριστήσω τους ε, ειδικού μας. Ήταν ενδιαφέρουσες οι συνεισφορές τους και πολλά ζητήματα έχουν αγερθεί. Εδώ έχουμε ζητήματα, ερωτηματικά και ανησυχίες που έχουν ακουστεί και σε επίπεδο συμβουλίου. Αυτό ήθελα να πω προ στιγμή, διότι δεν έχω προετοιμάσει κάτι για να απαντήσω σε ερωτήσεις των εμπειρογνωμόνων ή των βουλευτών. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις αντιδράσεις των εμπειρογνωμόνων και ίσως τότε να δευτερολογήσω. So, Mr. Καλά, ο κύριος Σούχα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πακ. Πρώτα απ' όλα για την ερώτηση στην οποία θέλετε να απαντήσω. Στο τέλος ή θέλετε να ακούσετε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τώρα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε στις ερωτήσεις και των εμπειρογνωμόνων και των συναδέλφων το, το θεώρησα καλύτερο να μιλήσετε πρώτα εσεί για να έχουν την ευκαιρία να αντιδράσουν σε αυτά που θα πείτε οι εμπειρογνώμονε. Εσάς θα σας ξαναδούμε τους επόμενους μήνες. Οι εμπειρογνώμονε είναι μόνο σήμερα εδώ. Λοιπόν, μόνο τώρα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μετά να απαντήσουν εκείνοι. Okay, thank you very much. Um, so first... Σας ευχαριστώ να ξεκινήσω με την απόκριση και απάντηση για την ε, Επίτροπο Βασιλείου. Δεν προσεκλήθη, δεν ε, υπήρχε αυτή η δυνατότητα σήμερα. Αλλιώ, οπωσδήποτε θα ήταν πολύ χαρούμενη να έρθει και μόλι υπευλήθηκε το πρόγραμμα ήδη από τον Νέμβριο του 2011, θυμάστε ότι είχε παρουσιάσει η ίδια το ε, όλο εγχείρημα εδώ στην Επιτροπή σα. Και να την υπερασπιστώ εδώ κάθε φορά που τη ζητούν οι Ευρωβουλευτέ να έρθει και να μιλήσει, το κάνει αυτό. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Then, uh, the, the, uh, Δεύτερο, ε, ε, το πρόγραμμα Creative Europe δεν αφορά την, ε, τον κλάδο, τον οικονομικό κλάδο της δημιουργίας. Εδώ υπάρχει παρανόηση δεν προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα για τον τομέα της δημιουργίας. Όχι, για τη δημιουργικότητα μιλάμε. Και εφόσον μιλάμε για τη δημιουργικότητα, ακριβώς αυτό που εννοούμε είναι αυτό που ανέφερε και ο Ράντου. Πάμε πίσω στον Αριστοτέλη. είναι αυτό το διαμάντι που μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθένα και στο πνεύμα του. Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατάλαβε επιτέλους. Κατάλαβε τη σημασία του ταλέντου και της δημιουργικότητας για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει και θεωρεί ότι η δημιουργικότητα που περνάει και τον πολιτισμό κατά την άποψή μας, μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και από την σκοπιά της έρευνας μέσα του Horizon 2020. Αυτές είναι οι βασικές στρατηγικές διεξόδου από την κρίση. Κατά αυτήν την έννοια είμαι περήφανο για την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει αυτό το μακρόπνο, το φιλόδοξο πρόγραμμα και αυτόν τον αυξημένο προπολογισμό για να το πρικοδοτήσει. Παρακαλώ καταλάβετε λοιπόν τι υπονοείται εδώ. Πίσω από το πρόγραμμα Creative Europe ακριβώ θέλουμε να οξύνουμε τα πνεύματα και να. Ε, έχουμε περισσότερο ήπια συναισθήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν οξύνια και ε, συναισθηματική θερμότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Αυτό θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης το 2020. Αυτό είναι το επίκεντρο και ο βασικός πρωταρχικός στόχος του προγράμματος. Δεν είναι οικονομικός και να μην είμαστε εδώ αφελείς. Βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, τα ανέφερε και ο Ράντου. Είναι πολύ καθοριστικό αυτό το μήνυμα. Βεβαίως ο πολιτισμός εδώ θέλει να καλύψει αυταξίες αλλά και την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη. Είναι πολιτικό λοιπόν το μήνυμα και αυτό το πολιτικό μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί με διαφορετικές νομικές βάσεις, διαφορετικά προγράμματα. Όχι, χρειάζεται ένα κοινό πρόγραμμα. Ενιαία θηρίδα θα την έλεγα. Όπως είπε και ο κύριος Καρούζο, έχουμε και τις ηλεκτρονικέ ταμπλέτες και τα εφή τηλέφωνα, αλλά δεν είναι μόνο οι ταινίε που περνάνε σε αυτέ τι συσκευέ. Και η μουσική και οι εικόνε και η λογοτεχνία και η πολιτιστική κληρονομιά, τα πάντα. Αυτές είναι οι προκλήσεις που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα καθοριστικά στοιχεία του πολιτιστικού τομέα συνενώνονται στο πρόγραμμά μας. Το είπαν και στις παρουσιάσεις οι εμπειρογνώμονες. Ε, ο ψηφιακό κόσμος σαφώς είναι αντικείμενο της αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σωστά, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σκέλος Κάτι που εμπεριέχεται και στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ποικιλία η πολιτιστική. Γι' αυτό έχουμε ως πρωταρχικό στόχο του προγράμματος να προωθήσουμε τη διαφορετικότητα. Πώς λοιπόν να λέμε ότι το πρόγραμμα αυτό προωθεί την οικονομία, εφόσον οι πρωταρχικοί στόχοι του είναι τόσο καλά εξισορροπημένοι. Αυτή λοιπόν είναι η βασική παρανόηση. Καταλάβετε ότι το πρόγραμμα Creative Europe είναι ένα έγγραφο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όχι το μόνο. Έχουμε ορίσει την πολιτική μας για τον πολιτισμό σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κρατη και τα γερμανικά κρατήδια και αυτό με την ατζέντα του 2007 για τον πολιτισμό. Αυτό το παρακολούθησαν και οι ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κρατη με την ε, μέθοδο ανοιχτού συντονισμού και όλα τα πονήματά μας, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από το 2007 μας οδηγούν προς το καινούριο εργαλείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Καταλάβετε όμως το πρόγραμμα Creative Europe είναι ένα εργαλείο στο φάσμα εργαλείων των πολιτιστικών που διαθέτουμε. Το είπαν και οι εμπειρογνώμονες. Έχουμε το IPI, έχουμε τα θέματα πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά δεν αποτελούν μέρη τη ε, δημιουργικής Ευρώπης. Έχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, τι κοινωνικέ εξελίξει το πρόγραμμα εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να τα απλουστεύουμε τόσο πολύ. Πρέπει να σεβαστούμε την αρχή τη επικούρικότητα επίση, αλλά και τι αρχέ ε, τη συμπληρωματικότητα. Δεν μπορούμε να προτείνουμε ένα πρόγραμμα που να επικεντρώνεται στον πολιτισμό και την εκπαίδευση μόνο. Πρέπει να ε, σκεφτούμε ότι έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Και δεν μπορούμε να προτείνουμε ένα θέμα για την ηθαγένεια λόγω χάρη, γιατί έχουμε ξεχωριστά προγράμματα γι' αυτό. Εδώ η πρωταρχική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προτείνει μέσα και εργαλεία που να είναι συμπληρωματικά. Γι' αυτό το συζητάμε. Καταλαβαίνουμε βεβαίω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίμερμαν ότι είναι προτεραιότητα ο πολιτισμός και η δημιουργία. Όμως το σκέλος αυτό και με το πρόγραμμα της διαβημάτισης καλύπτεται σε πολύ μεγάλο μέρος και θα καλύπτεται πλήρως από τα μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Γι' αυτό θέλουμε αυτό το καινοτόμο βήμα, την, ε, τον αλφαβητισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, της ψηφιακής ε, κοινωνίας. Πρέπει να δούμε πώς θα οθήσουμε το εκπαιδευτικό σκέλος σε ανάπτυξη. Το άνοιγμα των οριζόντων, πώς το κοινό θα εκτεθεί και σε νέες πολιτιστικές προκλήσεις και ρεθίσματα. Αλλά θέλουμε να το δούμε και από την εκπαιδευτική του σκοπιά όλο αυτό. Αυτό τώρα το κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό και το τι γίνεται με τις μικρότερες επιχειρήσεις και ενώσεις. Πρέπει εδώ να σοβαρευτούμε. Πρέπει να βασίσουμε τα επιχειρήματά μας σε πραγματικούς αριθμούς να σας πω τι γίνεται με τις μικρές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή 55% των οργανώσεων με λιγότερο από 11 εργαζομένους καλύπτονται από το τρέχον πρόγραμμα. Γιατί μιλάμε λοιπόν εδώ για τα μεγάλα προγράμματα. Πώς λέτε ότι δεν στηρίζουμε τις μικρές αλλά μόνο τις μεγάλες ενώσεις. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην προσέγγιση μας. Από το τρέχον πρόγραμμα στο μελλοντικό. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Ο μέσος όρος των επιδοτήσεων που μοιράζουμε είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Είμαστε λοιπόν, ε, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η Ευρώπη αποτελείται από μικρές και μικρότατες ενώσεις και επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει και το δημοσιονομικό μας μέσο. Αν δείτε το, το μέσο αυτό θα καταλάβετε ότι απευθύνεται μόνο σε μικρέ τέλο πάντων μικρομεσαίες επιχείρησει. Οι μεγάλες δεν θα έχουν πρόσβαση. Αυτά είναι τα στοιχεία που πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικά ε, για να γίνει σωστά αντιληπτό το πρόγραμμα. Ένα παράδειγμα, γιατί χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο μέσο. Το 2008 θα θυμάστε όλοι πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα με τις μικρές πολιτιστικές ε, ενώσεις στην Ευρώπη. Πολλά κράτη της Βαλτικής και κράτη της Κεντρικής Ευρώπης έχασαν τις πολιτιστικές τους ενώσεις, ε, επλήγησαν από τις δημοσιονομικές περικοπές. Εγώ λοιπόν συγκάλεσα μια συνεδρίαση του εκτελεστικού οργανισμού με τους συναδελφούς μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του είπα: ας δούμε μια άλλη νομική βάση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε βάση άλλη ε, νομική, άλλου άρθρου. Η γραφειοκρατική βέβαια προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί ήταν, ε, δεν μα επέτρεπε ευελιξία, νομική βάση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να υποστηρίξουμε αυτέ τι ενώσει με στοχοθετημένε δράσει πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε το Facebook, δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα. Το θυμάστε αυτό. Τώρα συντάσσουμε ένα κείμενο που θα πρέπει να πάει πέρα από το 2020. Εάν το πρόγραμμα λοιπόν λύγει το 2020, θα συνεχίσουμε τουλάχιστον για δύο-τρία χρόνια να υποστηρίζουμε τα ίδια προγράμματα. Προγραμματίζουμε λοιπόν για το απότερο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι προκλήσεις θα υπάρχουν στο μέλλον, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε στενά ώστε στο πνεύμα χάραξης πολιτικής και κατανόησης του τι προτείνουμε και για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον μικροσκοπικό προϋπολογισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σταγόνα στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι σαν μία βελόνα που χρησιμοποιεί βελονιστή για να θεραπεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πολιτιστικό δυναμικό που διαθέτει και για ένα καλύτερο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι. Ναι. Δεν είμαι τελείω σίγουρη εάν πήραμε απαντήσει στι ερωτήσει μα. Αλλά δεν θα πω τίποτα γιατί εγώ δεν ρώτησα τίποτα. Έχουμε χρόνο, να τα ξαναπούμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Μήπω να ακούσουμε του εμπειρογνώμονε μα πάλι. Ο κύριο Τσίμερμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έγιναν σε μένα ορισμένες ερωτήσεις και προτάσεις. Θα προσπαθήσω από το σύνολο να ξεχωρίσω ορισμένα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Όλοι οι πυρογνώμονες εδώ και οι ειδικοί ξέφυσαν τις ανησυχίες τους. Αν συγχωνευτούν αυτοί οι δύο τομείς της πολιτικής, τελικά μήπως πληγούν και οι δύο. Το θέμα δεν είναι να πληγεί το ένα πρόγραμμα και τα δύο τελικά θα βρουν τον πελά τους, ενδεχομένως. Και αυτό που ζητήσατε κυρία Πακ θα ήταν για μένα το ελάχιστο που θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Μια συγκεκριμένη εγγραφή με κονδύλια του προϋπολογισμού. Αν δεν μπορούμε έτσι και αλλιώς να διαχωρίσουμε τα δύο προγράμματα, τουλάχιστον να πούμε τι δίνουμε στο κάθε κονδύλι. Είμαστε βεβαίως υπέρ του να αυξηθεί η πρικοδότηση, έτσι κι αλλιώς. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Κάτι άλλο που με ανησυχεί εμένα είναι ότι το χρηματοδοτικό μέσο που εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο θολό. Ενδεχομένως στη συνέχεια να δημιουργηθούν εκεί δυσκολίες. Αν είναι και λιγότερα τα ποσά έτσι κι αλλιώς από εκείνα που επιθυμούμε όλοι μαζί. Γιατί εάν το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμοστεί ουσιαστικά θα ήταν ένα νέο στοιχείο του προγράμματος που δεν θα οδηγούσε σε ε, σαφή αύξηση των πόρων είτε του παλιού προγράμματος Μέντια είτε του παλιού προγράμματος για τον πολιτισμό και δεν θα είχε τη βάση του σε κανένα από τα δύο και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και προϋπόθεση. Θα πρέπει εκεί να ξεκαθαριστεί τι γίνεται και με το χρηματοδοτικό μέσο γιατί και αυτό είναι σαφές. Η κυρία Κάμερ Εβερτ ρώτησε για τις διάφορες δομές παροχής συμβουλών και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, τα σημεία επαφής για τον πολιτισμό, Cultural ε, contact points. Αυτό δεν είναι μόνο ένα σύμβουλος για το πώς θα κάνω την αίτηση για να πάρω επιδότηση για τον πολιτισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά τη διάρκεια των ετών αναπτύχθηκαν τελικά με μεγάλη επιτυχία σε ε, δομές ε, που βοηθούσαν τους καλλιτέχνες, γιατί πήγε ένας καλλιτέχνης μικρός και έλεγε ε, τι γίνεται στην Ευρώπη, με ποιον μπορώ να συνεργαστώ αν δεν είχαν εταίρους. Εκείνα τα σημεία επαφής τους έβρισκαν εταίρους, ε, δηλαδή ενεργά συμμετείχαν και βοηθούσαν τους καλλιτέχνες. αν θέλετε κάνανε και δουλειά συνεννόησης, επαφής των Ευρωπαίων μεταξύ τους, που υπερβαίνει κατά πολύ την τεχνική λειτουργία ενός γραφείου παροχής συμβουλών. Και βασικά ήταν καλλιτέχνες που απευθύνονται σε αυτούς και δεν είχαν ε, καθόλου εμπορικό προσανατολισμό προς την αγορά. Τώρα δεν ξέρω τι θα βγει από αυτή τη συγχώνευση. Αν συγχωνευτούν αυτά τα σημεία επαφή του πολιτισμού με τα λεγόμενα media desk. Βεβαίω κανεί μπορεί να φανταστεί ότι τελικά δεν θα αλλάξει τίποτα και όλα θα πάνε ωραία και καλά. Αλλά ανησυχούμε ότι μπορεί και να μην πάνε καλά. Αν πάει κάτι στραβά, τι γίνεται. Αν προκύψει μια κατάσταση που δεν ε, βοηθάει, εξού και η κριτική που εκφράζουμε πολύ. Και πολλοί ευρωβουλευτέ, ε, από ό,τι άκουσα. Αν είχε περιγραφεί καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια, δεν θα ανησυχούσαμε και θα ήμασταν πάρα πολύ ήρεμοι και νυφάλιοι. Και ο κύριος Σούχα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε μερικά στοιχεία, ε, τουλάχιστον με τις διαφορετικές έννοιες, χρειάζεται και διαφορετική αντιμετώπιση. Τι, η βιομηχανία της δημιουργίας είναι κάτι άλλο από την πρόθεση του πολιτισμού. Από τον ορισμό του τον ίδιο ένας κλάδος της βιομηχανίας και η βιομηχανία της δημιουργίας και ε, περιμένει να αποκομίσει κάποιο κέρδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προκύψει έτσι και αλλιώ το κέρδο, αλλά η ιδέα είναι ότι εγώ το κάνω γιατί είναι επάγγελμα, γιατί είναι εμπορική δραστηριότητα. Καλό είναι, θετικό, δεν το κατακρίνω και είμαι πάρα πολύ υπέρ. Και ο δικό μα φορέα θέλει να αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτό ο κλάδο, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο κάτι που δεν έχει σκοπό το κέρδο καθόλου. Και αυτό θα πρέπει να υπάρχει ως δυνατότητα. Δηλαδή να προωθούμε και ένα κλάδο που δεν θα αποφέρει κέρδος, που ακριβώς γι' αυτό του δίνουμε χρήματα, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η ύπαρξή του και γιατί δεν έχει οικονομικό όφελος, ούτε είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο προσανατολισμός του. Και για την πρωτοβουλία του 2020, όταν μου το λένε αυτό, αυτό με κάνει και ανησυχώ περισσότερο. Γιατί ακριβώς ε, εκεί αγωνιώ ότι θα πέσουμε περισσότερο στην οικονομία και λιγότερο στον πολιτισμό με το πρόγραμμα αυτό. Και αυτό ισχύει περισσότερο και προφανώς και για την εκπαίδευση, την πολιτιστική, που και ο Σούχα. Αυτό που είχαμε στη διαβίου μάθηση, από ό,τι ξέρουμε, δεν προβλέπει τίποτα για την πολιτιστική εκπαίδευση. Και θα πρέπει σε αυτό το πρόγραμμα του πολιτισμού να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Εγκαίρως λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να διορθωθούν ακόμα. Είναι όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα, είναι ρευστή η κατάσταση και καλό είναι που το συζητούμε αυτή τη στιγμή. Και ακριβώς είναι κρίσιμο, επειδή είναι λίγα τα χρήματα, να πούμε πού θέλουμε να στραφούμε αν θέλουμε να ενισχύσουμε και τα μίντια και τον πολιτισμό, να το ξεκαθαρίσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους. Αυτό ισχύει και για τη δική μας οργάνωση, το Γερμανικό Πολιτιστικό Συμβούλιο και να πούμε στη γερμανική κυβέρνηση ότι το πρόγραμμα είναι καλό και μην το πειράξετε και φροντίστε να βρείτε και τα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μιχαηλιάνο έχει το λόγο τώρα. Πώς προφέρετε το όνομά σας, Μιχαηλαιάνου? Euh, Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο πλευρές ε, που αναφέρθηκαν πολλές φορές αλλά δεν θα φτάσει ποτέ, θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, φοβόμουν πριν έρθω, αναρωτιόμουν μα θα με καταλάβουν, τελικά μιλάμε περίπου την ίδια γλώσσα. Και θα πω και θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα. Δεν πρέπει να έχουμε φλού στον προϋπολογισμό, δημοσιονομικά φλού, για πολλούς λόγους. Γιατί εμείς ε, οι δημιουργοί, ε, διανομι διανομής, παραγωγής, σκηνοθέτες, ηθοποίοι κτλ. Ε, πήραμε μία συνήθεια να δημιουργούμε μία πολιτιστική δυναμική γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο προπολογισμό, τον έχουμε βρει ποιο είναι και ξέρουμε ποιοι είναι και οι συνομιλητές μας. Και ακόμη και όταν υπάρχουν διαφορετικές χώρες μεταξύ τους με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία βοηθούν οι θεσμοί να μπορούμε να διαπιστώνουμε ποιοι είμαστε και το να συνομιλεί κανείς με έναν νέο ερχόμενο από ένα νέο τομέα που πάντα να συνεννοηθείς και πάνω να του εξηγήσει το έτοιμά σου κτλ. κτλ είναι ένα μπέρδεμα πραγματικά θα σκότωνε την όλη δυναμική, θα βάρινε στη δημιουργία και θα είχαμε δυσκολίες. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο ετέθη είναι πώς να μην εξαρτιόμαστε από την αγορά. Αυτή η περίφημη, αυτό το περίφημο ερώτημα που υπάρχει από πάντα, τι είναι η εμπορική τέχνη και τι είναι η καθαρή τέχνη. Εμείς στη Γαλλία καταφέραμε να βρούμε μία ισορροπία όπως τα πάντα στη ζωή και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λέμε ότι αυτοί που πρέπει να υποστηρίξουν την τέχνη είναι και οι δύο χρήστες της τέχνης, και ο ιδιωτικός τομέας και οι θεατές. Υπάρχει αυτό το ταμείο υποστήριξης, είναι μια χαζή ιδέα αν θέλετε. Όταν πάει κανείς και αγοράζει ένα εισιτήριο του στο σινεμά, το 18% από αυτό το εισιτήριο είτε είναι ένα αμερικάνικο φιλμ σαν τον Τιτανικό με 28 εκατομμύρια εισιτήρια πάει και χρηματοδοτεί το εθνικό σινεμά. Ό,τι λοιπόν έρχεται παρά από έξω που δεν είναι ευρωπαϊκό, πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά κάνει και έρχεται, υπέροχα, αλλά αυτό το έργο το οποίο θέλουμε απ' έξω να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πολιτιστική διαφορετικότητα, στη δημιουργία της. Στη Γαλλία γίνεται ένας ενδιαφέρον διάλογος και ισορροπημένος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συγχρηματοδοτούνται πολλές φορές τα φίλμα. και αυτό δημιουργεί διαφορετικότητα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναφέρατε για τις ποσοστώσεις. Φυσικά είμαστε σε ένα μοντέλο το οποίο δεν γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες, αλλά ε, εμείς έχουμε αυτή την ε, ψηφιακή επανάσταση με νέους που μπαίνουν στην αγορά και θέλουν να εκμεταλλευτούν την Ευρώπη και την αγορά της χωρίς να δώσουν τίποτα ως αντάλλαγμα. Θέλουν την, την διαφήμιση, θέλουν την προσοχή των Ευρωπαίων, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε κανόνες και ότι πολύ ωραία που έρχονται όλοι αυτοί οι σερβερ, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αναζήτησης, αλλά έχουμε όμως και μία αρχή ε, πολιτικής κουλτούρας που λέει ότι όποιος παίρνει πρέπει και να δίνει. Εντάξει, ανοίγει η αγορά, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξετε. Αυτό το οποίο πολλές φορές μπορεί και να σας έφτιαξε δηλαδή τον, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Γιατί βρίσκεται και στο δικό σας πετσί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν μπούμε σε μια δραματική φάση, δηλαδή στις τηλεοράσεις ίντερνετ, όπου έχουμε ε, τηλεοράσεις με ποσοστώσεις, τεφάν, τέντε και τα λοιπά, που συμβάλλουν στη δημιουργία έργων και τα πάνε μια χαρά οικονομικά. Και θα έχουμε λοιπόν σε αυτήν την τηλεόραση ίντερνετ αυτούς τους Ευρωπαίους χρήστες οι οποίοι συνεισφέρουν και αυτούς που δεν συνεισφέρουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Έτσι λοιπόν όσοι θέλουν το ευρωπαϊκό μάνα θα πρέπει να συμμετέχουν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χασμοντάλ, ο καθηγητής Χασμοντάλ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο για τις πολύτιμες συνεισφορές τους. Κύριε Καβαντά, δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσει ο κύριος Χέσμονταλ. Να ξεκινήσω με την κυρία με την παρατήρηση της κυρίας Τρούπελ κατά πόσο είναι θεμητό να συνεχίζεται η χρηματοδότηση για τις τέχνες και την ψυχαγωγία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς να πετύχουμε αύξηση σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Καταλαβαίνω γιατί τίθενται οικονομικοί στόχοι, ακόμα και σε τέτοιου καιρού, για να μπορέσει κανεί να αιτιολογήσει τη χρηματοδότηση του πολιτισμού και της τέχνης, αλλά υπάρχει και το ανάλογο κόστος και το εντοπίσατε κι εσείς. Ενδεχόμενη υποβάθμιση αυτών των πολύτιμων μορφών ανθρώπινης έκφρασης σε απλές μετρήσιμες δραστηριότητες. Για να συνεχιστούν λοιπόν οι επιδοτήσεις θα πρέπει να, χρησιμοποιηθούν τα επιχειρήματα των οικονομολόγων κατά των οικονομικίστικων απόψεων. Εξήγησα προηγουμένως ότι υπάρχουν επαλαμβανόμενα χαρακτηριστικά στην ε, πολιτιστική παραγωγή και οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν, στους, ε, δεν επιτρέπουν να ευδοκιμήσουν τα πολιτιστικά αγαθά εκεί. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι παρατηρήσει του κυρίου Σκουρία. Πώς θα προστατεύσουμε τον πολιτιστικό τομέα στην πράξη. Πώς θα προστατεύσουμε τις μικρότερες ομάδες και ενώσει, Πιστεύω ότι το θέμα των desk των γραφείων είναι πολύ σημαντικό. Τα media desk που λειτουργήσαν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και κατά πόσο μπορούν να συγχωνευθούν. Δεν είμαι αντίθετος. Απλώς έλεγα ότι πρέπει να ορίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την ιδιαίτερη αντίληψη των ιδιαίτερων οτροπιών που μπορεί να, γίνει να προκύψει με την συγχώνευση των ε, media desk. Επίσης μπορεί να υπάρξει ε, κάποια κάλυψη του εμπορικού σκέλους με το μη κερδοσκοπικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ομάδα, ομάδα που να συνδυάζει διαφορετικές εμπειρογνωμοσύνες και γνώσεις. Νομίζω ότι απαντώ έτσι και στο ερώτημα της κυρίας Κάμερβερτ σύντομα να στραφώ και στις παρατηρήσεις του εκπροσώπου της Επιτροπής. Και ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά τη δημιουργικότητα, το και έχει την, ε, τον κλάδο της βιομηχανικής ε, δημιουργίας στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Μεγάλο μέρος του προγράμματος δεν αφορά ακριβώς τον κλάδο της δημιουργίας. Αλλά αυτό που ήθελα να πω με την παρουσίασή μου ότι η συμπερίληψη ρητορικών επιχειρημάτων, όπως η θέρμανση των συναισθημάτων και η όξυνση του νου, μας θυμίζει το τι συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες για πολλές εθνικές πολιτικές για τον πολιτισμό. Και αυτές, αυτοί οι απόέχοι θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Κάτι που έγινε σε μερικές χώρες, όπως και στην Πρετανία, είναι ότι τα επιχειρήματα υπέρ της δημιουργικότητας και την οικονομική της αξία χρησιμοποιήθηκαν τελικά για περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά πολλοί από τους συμμετέχοντες στον τομέα της ε, δημιουργίας που δεν είναι κερδοσκοπικός βρέθηκαν να πολιορκούνται από ένα σωρό απαιτήσει και επιταγές που τελικά ε, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν αυτό που θέλαν ε, για να προσφέρουν ε, στην έκφραση της ανθρώπινης κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά μας είπε ότι το πρόγραμμα για τα πολιτιστικά έχει στηρίξει κάποιε μικρότερε οργανώσει. 55% τη χρηματοδότηση δηλαδή πηγαίνει σε επιχειρήσει ή ενώσει με λιγότερου από 11 εργαζομένου. Αυτό είναι αξιέπαινο. Όμω, το θέμα είναι κατά πόσον αυτόν θα εξακολουθήσει. Θα υπάρχει επαρκή προστασία. Θα, υπάρχει, θα υπάρχουν επαρκή εχέγγυα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Διότι εξ όσων καταλαβαίνω, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση και στο σκέλος του πολιτισμού και στο σκέλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά οι μη κερδοσκοπικές ε, οργανώσεις δεν θα έχουν καμία πρόσβαση ή τέλος πάντων περιορισμένοι στο συνολικό προπολογισμό. Εκεί γίνονται ερωτήματα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ναι, φαίνεται να μιλάμε εδώ κατεξοχήν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της δημιουργίας, της ψυχακογίας, πίνουν να είναι πανίσχυρες λόγω της ανεπίσημης χρηματοδότησης των συσχετισμών που έχουν με τις ε, πολυεθνικές. Αυτό τους δίνει δυνατότητα άσκησης πίεσης. Και πιστέψτε με, στον τομέα της ψυχαγωγίας Ακριβώ επειδή υπάρχουν τέτοιε μάχε με τα δικαιώματα τα πνευματικά και τα δικαιώματα πνευματικού δημιουργού τα τελευταία 20 χρόνια, είναι τεράστια δυνατότητα άσκηση πίεση. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ακόμα και με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορεί να ε, υπάρξει κατακράτηση των κονδυλίων και να καταλήξουν τελικά σε αυτά τα χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καρόσο για να κλείσει. Ο κύριος Καρόσο εμπειρογνώμων και αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πάκ. Εγώ θέλω να απαντήσω στο σχόλιο της κυρίας Κώστα σχετικά με το κατά πόσο ή όχι θα πρέπει να πληρώνονται οι πλατφόρμες, όπως γίνεται και στη Γαλλία. Το θέμα των νέων γιγάντων της, παρα... της διανομής είναι ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεφύγουν από τη φορολόγηση όπως συμβαίνει με το Google εξάλλου που δεν εγκαταστάθηκε στη Γαλλία αλλά θα πάει στην Ιρλανδία. Και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ε, διανομέας που θα πάει στο Λουξεμβούργο και όχι στη Γαλλία για να ξεφύγει από τη γαλλική νομοθεσία που επιβάλλει την καταβολή ενός ποσοστού ε, του κύκλου εργασιών στην ανεξάρτητη παραγωγή. Εγώ δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο γιατί το, τα είπαν οι συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι από τις τοποθετήσεις των εμπειρογνωμόνων στον πολιτισμό, από την τοποθέτηση του Ράντου, αλλά και στην ρεαλιστική τοποθέτηση του κυρίου Καβαντά, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική βούληση έστω και κάτω από την ίδια ομπρέλα να παραμείνουν τα δύο προγράμματα ανεξάρτητα και αυτόνομα και οικονομικά και διοικητικά. Μπορούν να υπάρξουν συνέργειες, ε, είναι χρήσιμες και απαραίτητες για τα προγράμματα. Σκέφτομαι εδώ το cross media, δεν είναι μόνο ε, ακουστικό, μπορεί να περάσει και στο offline όπου το, το όπου με πειράματα που έγιναν στην Σουηδία βλέπουμε ότι offline μπορεί να λειτουργήσει και για το θέατρο, το χορό. Ίσως θα χρειαζόμασταν ε, ένα καλύτερο ορισμό και περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονές μας. Θεωρώ ότι μας έχετε υποστηρίξει πολύ στη προσπάθειά μας. Ε, σημειώσαμε πολλά και φιλοσοφικά και χαίρομαι που χαρήκατε και που εκπλαγήκατε ε, που σκεφτόμαστε ε, το ίδιο με εσά. Εμείς είμαστε καλύτεροι από τη φήμη μας, ανέκαθεν, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει, αυτό είναι το θέμα. Θα ήθελα να συνοψίσω πάρα πολύ σύντομα και να πω και προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πολύ ωραία τα λόγια αυτά που είπατε αλλά ουσία πουθενά. Δεν μας απαντήσατε για τις αγωνίες και τους φόβους μας και είπατε πολλά από αυτά που φοβόμασταν για τον ορίζοντα 20. δεν είναι αυτό το θέμα εδώ ορίζον του 2020. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Προφανώ έχει επιπτώσει σε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα και σε άλλου τομεί. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Αλλά το κρίσιμο και το ουσιώδε δεν είναι το ορίζον 2020 και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένο και ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό να το βλέπει μόνο υπό το πρίσμα του ορίζον 2020. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ ισχνή απάντηση. Όλοι οι πυρογνώμονε είπαν ότι πολιτιστική πολιτική και ο πολιτισμός είναι δίκτυα. Να δικτυώνονται οι καλλιτέχνες, τα μεμονωμένα σχέδια, έργα. Αυτό δεν το αναφέρατε. Μας είπατε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικονομία είναι, επιχειρήσεις είναι. Εντάξει, να στηρίξουμε τις μικρές, αλλά τώρα το λέω προσωπικά. Δεν είμαι υπέρ του να λέμε στο κείμενο, όπως το λέτε, expresses verbis, ότι, πώς τα λένε αυτά τα video games, τα, παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά. Σιγά, αυτή η αγορά μπορεί από μόνη της να ανθίσει, που ανθεί και να πλουτίσει. Δεν χρειάζεται τη δική μας υποστήριξη. Έτσι κι αλλιώς ε, είχα εκνευριστεί και στην παρουσίαση και τα έχω ξαναπεί αυτά. Αυτά που μας είπατε πιστεύω ότι δεν ήταν ακριβή, ούτε συγκεκριμένα, ούτε μπόρεσαν οι επιρογνώμονες να βρουν απάντηση στα όσα στυλίτευαν. Εμείς δεν θέλουμε λόγια να μας χαϊδεύουν τα αυτιά, θέλουμε ακρίβεια, σαφήνεια και εγγραφή των κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε επίσης συγκεκριμένη συζήτηση για τη χρηματοδότηση. Αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων που μας χρειάζεται για το χρηματοδοτικό μέσο να το χειριστούμε, που εγώ πιστεύω έτσι εκ πρώτης όψης ότι μπορεί να δουλέψει, αλλά αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων είναι ένα τμήμα του μικρού μας προϋπολογισμού ήδη από την αρχή αφαιρεί ένα τμήμα που θα θέλαμε να έχουμε να το χρησιμοποιούμε αλλού. Και αν δεν χρησιμοποιηθεί, τι θα γίνουν τα λεφτά αυτά του Ταμείου Εγγύσεων. Θα γυρίσουν πίσω γενικά στα κράτη-μέλη, στους καθαρούς συνεισφορείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον πολιτισμό, γενικά έχουμε την ερώτηση αυτή. Και στην παιδεία, ας πούμε. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, η δυνατότητα στήριξης των δανείων Καταρχήν, το καλωσορίζουμε, αλλά πώς θα λειτουργήσει. Θέλει μεγάλη συζήτηση και αυτό. Μετά έγινε ερώτηση αν θα πρέπει να συνενωθούν το Media Desk και τα σημεία επαφής ε, για τον πολιτισμό. Εδώ υπάρχουν υπέρ και κατά. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικοί συνομιλητές αυτές οι υπηρεσίες. Και εγώ δεν θέλω να ε, υπονομευτεί ε, είτε ο ένας είτε ο άλλος από τη συγχώνευση. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να αλλάξει η δομή τους, αλλά να συγχωνευτούν και ότι θα έχουν και οικονομική συνέργεια και συνέργεια γενικότερα, δεν ξέρω. Τολμώ να το αμφισβητήσω. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι ομάδες οι μονάδες επαφής για τα πολιτιστικά προγράμματα συγγνώμη, βοήθησε πάρα πολύ τους καλλιτέχνες αν συγχωνευτούν και αυτά. Εντάξει, δεν θα το κλείσουμε, δεν θα το ολοκληρώσουμε σήμερα εδώ ότι είναι οριστικά αυτά που λέμε. Και κάτι άλλο που το έχουμε ξανασυζητήσει. Στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί κανείς να επιλέξει πού θα πάει για να εξοικονομήσει χρήματα από τον πολιτισμό. Αν θα πάει στο Λουξεμβούργο ή στην Ιρλανδία, α πούμε, μια εταιρεία. Αυτό πια δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Εδώ θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση και η ευρωπαϊκή αγορά εδώ να γίνει ενιαία αγορά. Τώρα βέβαια έχουμε το πρόβλημα ότι η φορολογική πολιτική δεν είναι εναρμονισμένη, αλλά σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στις κυβερνήσεις στην Ιρλανδία και στο Λουξεμβούργο προς όφελος του πολιτισμού αυτό να μην το επιτρέπουν. Ναι. Εντάξει, η αισιοδοξία είναι καλό πράγμα. Και θα πρέπει να πιστεύουμε στην καλή διάσταση του ανθρώπου και του πολιτικού εν γέννη, για να προχωρήσουμε. Πάντως να το θέσουμε αυτό το ζήτημα. Τι μάθαμε σήμερα λοιπόν. Όλοι οι εμπειρογνώμονες και εκείνοι που εκπροσωπούν τα μέσα, τα οπτικοακουστικά, ενδιαφέρονται να προωθεί και η μη κερδοσκοπική διάσταση ε, του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες, να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μαζί τους και να πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της μικρής κατά τα άλλα πίτας. Για το συνολικό ποσό και πάλι δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι, αλλά χαίρομαι πολύ που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξηθεί κατά 37%. Αυτό το έχει δηλώσει. Και αν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι το συνολικό ποσό, θα πρέπει να καθίσουμε τα τρία θεσμικά όργανα και να πούμε ότι θα αυξηθεί κατά 37% από αυτό που είχαμε. Το ελάχιστο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ανοίξει η μύτη ούτε στα διαρθρωτικά ταμεία, ούτε στις γεωργικές δαπάνες, αν πάρουμε ένα μικρό κονδύλι. Και αυτό πραγματικά, ξέρετε, είναι η ψυχή της Ευρώπης. Ευχαριστώ λοιπόν εξ ονόματος όλων των συναδέλφων και σας εύχομαι να παραμείνουμε σε επαφή για να έχουμε τελικά ένα καλό πρόγραμμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τιτανική Προεδρία. Και την Κυπριακή, την επόμενη. Γιατί όλα αυτά θα τα δούμε και στην αρχή του επομένου α, που θα είναι η Κυρλανδία, Εκεί θα τους τα πούμε τα φορολογικά, θα τις τα τρίψουμε στα μούτρα. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη της ακρόασης. Ευχαριστώ πάλι. Και θα σας χειροκροτήσουμε πολύ θερμά. Σημείο 11. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Όχι 11, 14 Δεν διαφωνεί κανείς. 15 διάφορα, έχετε κανένα διάφορο. Όχι, 16 προσεχή συνεδρίες 29 Μαΐου το πρωί στις 9 και το απόγευμα στις 3. Δεν είναι δύο μισές μέρες, μία μέρα απόγευμα και άλλη το πρωί. Όχι, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεδρίες, χαίρετε.